Um, Έλεγα λοιπόν καλό απόγευμα, λέει ο πρόεδρος. Μας λείπουν κάποια μέλη. Ο κύριος Αλάρντ ε, διεκόπη πριν τη διακοπή για το γεύμα και άλλα μέλη δεν είχαν καν την ευκαιρία να υποβάλουν το ερώτημά τους. Ο κύριος Αλάρντ έλεγε ότι δεν είναι σαφές για τα νέα μέλη πώς εκδηλώνουν ενδιαφέρον να λάβουν το λόγο ή να κάνουν μια ερώτηση. Και έχοντας συμπληρώσει 15 χρόνια εδώ μέσα, ε, συνηθίζει κανείς τη διαδικασία, λέει ο Πρόεδρος. Λέω λοιπόν, όταν ξεκινάμε ένα σημείο, ένα επόμενο σημείο στη διάταξη και το ανοίγουμε, από εκεί πέρα μπορείτε απλώς να σηκώνετε την καρτέλα σας ώστε η γραμματεία να σημειώνει ότι θέλετε να προσθεθείτε στον κατάλογο των ομιλητών. Η κανονική διαδικασία είναι ότι ο πρόεδρος συνήθως δίνει στους συντενιστές πρώτα το λόγο και μετά πάμε οι συγητές και συντονιστές όπως αντιλαμβάνεστε έχουν ειδική μεταχείριση αλλά από εκεί και πέρα κατά προτεραιότητα που έχετε ζητήσει. και αν μακρηγορήσουμε υπερβολικά, τότε ο πρόεδρος μπορεί να πει ότι κλείνουμε τον κατάλογο. Άρα, αν σας ενδιαφέρει το θέμα, να ζητάτε το λόγο νωρίς. Μετά την εισαγωγή αυτή, θα πάω στον κανονισμό ελέγχων, π.χ. τώρα αν θέλετε να ζητήσετε λόγο μετά να το εκδηλώσετε ήδη. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν υπό την προηγούμενη θητεία προφανώς. Προκατακτική δουλειά έγινε από τους σοσιαλιστές. Ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν ξέρω αν το SND ονόμασε τον συγητή τους. Η κυρία Βάιτς τώρα εκπροσωπεί την Κομισιόν. Θα την καλούσα να μας κάνει μια εισαγωγή στον κανονισμό ελέγχων. Η πλειοψηφία των μελών μάλλον δεν έχει διαβάσει τον κανονισμό. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάποιες βασικές αρχές, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλους, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά σήμερα να σας παρουσιάσουμε με συνεπέστερο τρόπο ελπίζω τον κανονισμό των ελέγχων, ο οποίο την επανεξέτασή του δηλαδή, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την πρόταση της Κομισιόν. Προκειμένου να εξηγήσω, θα έχουμε μία παρουσίαση PowerPoint, λόγω των οποίων και κάθομαι εδώ που κάθομαι. Θα είναι παρουσίαση και από μένα και από τη Φραντσέσκα και καθότι πρώτη φορά μας βλέπετε οι περισσότεροι. Βερόνικα Φάιτς, διευθύντρια στη Μάρε για την ΚΑΠ συμπεριλαμβανομένου του EMFF, του κανονισμού ελέγχων και την υλοποίηση για Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Η Φρανσέσκα Ρένα, επικεφαλής των ελέγχων και επιθεωρήσεων στη Μάρε. Πάμε στην πρώτη διαφάνεια. η οποία είναι μια γραφική παρουσίαση που σας δείχνει οπτικά ότι η έλεγχη και η επιτήρηση είναι η ραχοκοκαλιά, λέει η μιλήτρια της κοινή πολιτικής αλίας, των βασικών αρχών δηλαδή του κανονισμού, στο μέσον βλέπετε ότι οι αρχές και οι στόχοι υλοποιούνται μέσω δυνατοτήτων πολιετών σχεδίων διαχείρισης, τεχνικών μέτρων και τα μέτρα αυτά προστασίας ε, βασίζονται σε επιστημονικές συμβουλές. Δεδομένα δηλαδή και επιστημονικά, αλλά και που προκύπτουν από την επιτήρηση και τον έλεγχο του στόλου. Από την ελευτική δηλαδή προσπάθεια. Μπορεί να έχει κανείς τα καλύτερα στον κόσμο μέτρα προστασίας, αλλά δεν θα λειτουργήσουν εφόσον δεν υλοποιηθούν και δεν ελεγχθεί σωστά η εκτέλεσή τους. Θα έχουν λοιπόν πραγματικά θετικό αντίκτυπο και ευκταίο αντίκτυπο εφόσον υλοποιηθούν από τον κλάδο και ελεγχθούν επαρκώς, συνολικά. Ο στόχος του συστήματος ελέγχων είναι να συνεισφέρει στους στόχους της ε, ΚΑΠ, δηλαδή να εξασφαλίσει βιώσιμο απόθεμα πόρων και αλληλευτικής δραστηριότητας παρακολουθώντας τις ε, αλλιευτικές ε, προσπάθειες, τις δραστηριότητες, ποιος αλλιεύει, πού, πόσο και πότε. Αυτή είναι σημαντική διάσταση του στήματος ελέγχου, γιατί παρέχει κρίσιμα στοιχεία για τους υπεύθυνου διαχείρισης, ώστε να προβούν σε επαρκή κατάλληλη διαχείριση του αποθέματος. Και χρειάζονται επίκαιρες και ακριβείς αξιολογήσεις του αποθέματος. Η δεύτερη δέσμη δράσεων είναι να έχουμε μηχανισμούς που θα εξασφαλίζουν ότι οι αλληλείς συμμορφούνται προς τους κανόνες και αποτρέπουν παράνομη δραστηριότητα. Δηλαδή χρειαζόμαστε κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Η τρίτη δέσμη είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της ε, παράνομης λαθρείας και άναρχης αλίας, δηλαδή της γνωστής IUU. Αργότερα έχετε αντίστοιχο σημείο στη διάταξη, δεν θα επεκταθώ επ' αυτού. Η φυστάμενη νομική βάση ποια είναι. Έχουμε τέσσερις συμπληρωματικούς πυλώνες. Πάνω αριστερά έχετε τον κανονισμό ελέγχου του 2009 που τότε ήταν πολύ σημαντική επικαιροποίηση όλων των κανόνων. Στα δεξιά έχουμε τον κανονισμό για την άναρχη από το 2008. Κάτω αριστερά ε, έχετε τον ε, συστατικό κανονισμό της ΕΦΚΑ, δηλαδή τους συστατικούς κανόνες για τον οργανισμό ελέγχου, οργανισμός δηλαδή που συντονίζει τις προσπάθειες ελέγχου των κρατών μελών και τέλος βέβαια την βιώσιμη διαχείριση του εξωτερικού στόχου, ε, στόλου. Με συγχωρείτε. Έχουμε επανεξετάσει το 2017 και εδώ μιλούμε για τη διαχείριση του στόλου μας σε εξωτερικά ύδατα ή εξωτερικούς στόλους στα δικά μας ύδατα. Έχουμε μια σειρά από άλλα νομοθετικά μέτρα με μέτρα ελέγχου για τον κανονισμό για τη Μεσόγειο, τον Βεθυπελαγικό διατάξει ελέγχου και επίσης άλλες διατάξει ελέγχου που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες. Πρόκειται λοιπόν για ένα εκτεταμένο νομικό πλαίσιο, όπως κάθε νομοθετικό πλαίσιο όμως πρέπει να ξανακοιτούμε από καιρούς καιρών την αποτελεσματικότητά του μέσω ενδελεχούς αξιολόγησης. Αυτό έκανε η Κομισιόν του 2017 και αυτό έκανε και το ελεγκτικό συνέδριο την ίδια χρονιά το 2017. Και ως εκ τούτου το συνέδριο εξέδωσε έκθεση με τίτλο «Νέοι έλεγχοι για την ΚΑΠ απαιτούνται νέοι έλεγχοι». Απευθυνόμενο στον οργανισμό, το κοινοβούλιο εδώ υιοθέτησε ψήφισμα το 16 ώστε να είναι ομοιόμορφη η έλεγχη γελιευτική στην Ένωση. Έχουμε λοιπόν διάφορε αξιολογήσει και τα τελευταία χρόνια και αυτό που προκύπτει από όλες αυτές τις αξιολογήσει και επανεξετάσεις είναι ότι συγκλίνει, συγκλίνουν όλες, όλα τα πορίσματα προς την άποψη ότι αυτή τη στιγμή το πλαίσιο δεν είναι απόλυτα επαρκές και οδηγούμαστε σε τέσσερις περιοχές όπου απαιτούνται βελτιώσεις. Καταρχά, η συλλογή δεδομένων αλληλεία, ειδικά μικρή κλίμακα και βιοτεχνική κλίμακα αλληλεία, είναι ανεπαρκή τα δεδομένα αυτά. Ω εκ τούτου, έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία τα στοιχεία αυτά τα δεν είναι πλήρη, δεν είναι απολύτως διαθέσιμα και δεν είναι απολύτω αξιόπιστα. Η δεύτερη περιοχή προς βελτίωση είναι η επιβολή. Η αξιολόγηση ξεκάθαρα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πολύ άνηση επιβολή, υλοποίηση δηλαδή από πλευρά των κρατών μελών και επομένως άνισο πεδίο παιχνιδιού. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορα όρια, μάλλον διάφορα επίπεδα κύρωσης για την ίδια παράβαση σε διαφορετικά κράτη-μέλη. άνιση κανόνες δηλαδή. Επίσης, το σύστημα ελέγχων δεν ευθυγραμμίζεται με τη νέα κοινή αντιληφτική πολιτική από το 2014, ιδιαίτερα δε ως προς τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Και ο Γενικός Διευθυντής Ματσάδο σας μίλησε συγκεκριμένα για αυτό. Η τέταρτη βελτίωση είναι η υπερβολική περιπλοκότητα των υφιστάμενων κανόνων με πολλές και διάφορες εξαιρέσεις δυσκόλως ελέγξιμες και έλλειψη αφήνειας διαφόρων άλλων διατάξεων. Υπό το φως λοιπόν του συνόλου αυτούς συστάσεων και αξιολογήσεων ήταν σαφές για μας στην Κομισιόν ότι το να μην αναλάβουμε δράση δεν ήταν δυνατό ως επιλογή. Επί τη βάση αξιολόγηση αντικτύπου πλήρη, υιοθετήθηκε μια πρόταση το τέλος Μαΐου του 18, έκτοτε συζητείται από τους συνομοθέτες. Και τι κάνει η πρόταση αυτή, για να είμαστε σαφείς, δεν μιλούμε για αναστολή, ανάκληση του υφιστάμενου στήματος. Μιλάμε για τροποποίηση του υφιστάμενου στήματος στις περιοχές εκείνες που κρίναμε ότι ήταν απαραίτητο. Και αφορά αυτό σε τρεις βασικούς κανονισμούς, εκείνων των ελέγχων, τον στατικό της ΕΦΚΑ και της IUU με μικρέ τροποποίησεις και σε άλλου κανονισμού όπως εκείνη του Μεσογείου και τη βαλτική ε, το σχέδιο διαχείριση. Αυτό είναι το πλαίσιο της επανεξέτασης του συστήματο ελέγχων. Η Φραντσέσκα επίση σύντομα ελπίζω θα σας ε, παρουσιάσει το περιεχόμενο όλων αυτών των τροπολογιών. Uh, Καλησπέρα σα. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τώρα το περιεχόμενο της πρότασης εστιάζοντας στις πιο σημαντικές ε, τροποποιήσεις που έγιναν στις διατάξεις και τις έχουμε κατηγοριοποιήσει εδώ στους ε, κανόνε επιβολή τη νομοθεσία, διαθεσιμότητα των δεδομένων, ζητήματα όπου θα πρέπει να γεφυρώσουμε το ε, κενό που υπάρχει μεταξύ αυτών των ε, κανονισμών ε, με την κοινή αλληλευτική πολιτική, τι αυξημένε συνέργεια και επίση ε, τι αλλαγέ που θα γίνουν στον κανονισμό σε ό,τι αφορά την ίδρυση τη ΕΦΚΑ και τον κανονισμό σε σχέση με την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία. Κάτι που θα πρέπει να πούμε ευθύ εξ αρχή είναι ότι με αυτή την πρόταση προσπαθούμε να ε, διευκρινίσουμε τους υφιστάμενους κανόνες και να πλουστεύσουμε το κανονιστικό πλαίσιο. Ε, βέβαια αυτό είναι δύσκολο καθώς επόκειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης ε, προσπαθήσαμε εδώ να καταργήσουμε με την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων κάθε είδους σε έγγραφη μορφή, σε έντυπη μορφή. Προσπαθήσαμε δηλαδή να κινηθούμε πιο πολύ προς την ψηφιοποίηση αλλά και να ευθυγραμμιστούμε με τα όσα προβλέπει ε, η Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά λοιπόν το κομμάτι τη επιβολή τη νομοθεσία, θα εστιάσω ιδιαίτερα στι κυρώσει. Εδώ λοιπόν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία και μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προτείνουμε είναι να συνδυάσουμε όλες τις διατάξεις οι οποίες αφορούν κυρώσεις και παραβάσεις σε έναν κοινό κανονισμό που θα είναι ακριβώς αυτός ο μελλοντικό κανονισμός ελέγχου στην Αλία. Δηλαδή, ε, οι υφιστάμενε ε, σχετικέ διατάξει σε ό,τι αφορά κυρώσει που περιλαμβάνονται αυτήν τη στιγμή στον κανονισμό για την αλληλεία IUU θα περιλαμβάνονται στο μέλλον στον κανονισμό για του ελέγχου. Επίση, προτείνουμε να υπάρχει μια ενημερωμένη λίστα, σε ενημερωμένο κατάλογο ω προ το τι αποτελούν αυτέ αυτές καθ' αυτές ε, σημαντικές ή σοβαρέ παραβάσει, Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιε οι οποίε θεωρούνται σοβαρέ, ενώ άλλε θεωρούνται σοβαρέ κατά τη διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτου μέλου. Άρα λοιπόν ο τρόπο με τον οποίο γίνεται η ερμηνεία αυτών των παραβάσεων, σοβαρέ ή όχι, εξαρτάται από το κάθε κράτο μέλο. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνουμε να έχουμε πιο εναρμονισμένα κριτήρια έτσι ώστε να θεωρούνται και ε, περαιτέρω ε, παραβάσεις οι οποίε αφορούν ακριβώ του κανόνε κοινή αλληλευτικής πολιτικής ω σοβαρέ ή μη σοβαρέ. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να έχουμε ένα πιο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο στο σύνολο του τομέα. Επίση, προβλέπουμε μια σειρά από υποχρεωτικές ε, διοικητικέ κυρώσει και ελάχιστα επίπεδα ε, προστήμων σε ό,τι αφορά τι σοβαρέ παραβάσει, πράγματα τα οποία δεν ίσια μέχρι σήμερα. Ε, και αυτό ισχύει γιατί μέχρι στιγμή, επειδή ακριβώ η αντιμετώπιση των παραβάσεων περνάει μέσα από το ποινικό σύστημα συχνά έχουμε μεγάλε καθυστερήσει στην όλη διαδικασία ε, πολλαπλών ετών. Οπότε λοιπόν θέλουμε να έχουμε την επιβολή τέτοιου είδου κυρώσεων και προστήμων και ταυτόχρονα παρακολούθηση τη διαδικασία και τρέξιμο τη διαδικασία μέσα του ποινικού συστήματο των κρατών μελών. Από εκεί και μετά θέλουμε την επιβολή ε, άμεσων μέτρων επιβολή τη νομοθεσία σε περίπτωση που εντοπίζεται μια ε, παράβαση και επίση προσπαθούμε να έχουμε πλέον μια ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τι κυρώσει και τι παραβάσει. Ε, δεύτερο σημαντικό κομμάτι των αλλαγών αφορά στη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την διαθεσιμότητα αλλά και την ποιότητα των δεδομένων σε ό,τι αφορά όλα τα είδη σκαφών. Ξεκινάμε δηλαδή καταρχήν με μικρού μεγέθους ε, σκάφη, δηλαδή μικρότερα των 12 μέτρων, για τα οποία μέχρι στιγμής ισχύουν μια σειρά από εξαιρέσεις από την νομοθεσία. Για παράδειγμα, έως 10 μέτρων ε, ε, μήκος δεν έχουν την υποχρέωση τη σήμερα ημέρα να αναφέρονται σε κανενός είδους αλλιεύματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν για αυτά τα σκάφη προβλέπεται ε, υποχρεωτική ανείχνευση, δηλαδή να παρακολουθείτε ε, η θέση του σκάφους και επίσης υποβολή εκθέσεων, δηλαδή αναφορές σε ό,τι αφορά τα αλλιεύματα αυτών των σκαφών, με βάση μία σειρά από απλά εργαλεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό για ακριβώς αυτά τα μικρά ε, σκάφη. Αντί δηλαδή για τα πιο περίπλοκα και βαριά εντό εισαγωγικών συστήματα που είναι πιο ενδεδειγμένα για μεγαλύτερα σκάφη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σκάφη ε, μεγαλύτερα από 12 ε, μέτρα, έχουμε ε, εξαιρέσει αυτά από τις υφιστάμενες αποκλήσεις που ίσχυαν για, για παράδειγμα σκάφη ως των 15 μέτρων σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την παρακολούθησή τους, την αντίγνευσή τους. Και πάλι δηλαδή εδώ ισχύει πλέον ότι δεν θα υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις και θα πέρα από την παρακολούθηση θα πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονικά τις αναφορές τους. Επίσης, Έχουμε κάνει μια αναθεώρηση του άρθρου ε, σε ό,τι αφορά την ερασιτεχνική αλληλεία. Το εν λόγω άρθρο, η εν λόγω διάταξη, ε, δεν είναι καθόλου ισχυρή τη σήμερα ημέρα. Δηλαδή, ε, δεν εξασφαλίζεται ο έλεγχο ε, ο έλεγχο τη επιβολή τη. Οπότε, επειδή ακριβώ δεν υπάρχουν και συστήματα διοδότηση συχνά, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο και ούτε γνωρίζουμε το ποια είναι τα αλλιεύματα αυτών των ερασιτεχνικών αλλιέων. Άρα, λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει ένα σύστημα ε, εγγραφή σε μητρό και αδειοδότηση στα κράτη-μέλη, χωρί ωστόσο να ορίζουμε πώ θα ισχύει, πώ θα λειτουργεί αυτό το σύστημα σε κάθε κράτο μέλο. Και επίση, ε, προβλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα συλλογή δεδομένων και καταχώρηση των δεδομένων σε ό,τι αφορά όλα τα ίδια αλλιευμάτων σε ό,τι αφορά τα είδη για τα οποία υπάρχουν ε, μέτρα συντήρησης των αποθεμάτων σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, προτείνουμε τη δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών, όπως δηλαδή αυτό προβλέπεται τη σήμερα ημέρα για τα μικρού μεγέθους σκάφη. Σε ό,τι αφορά πάντα το ζήτημα των δεδομένων, έχουμε καταργήσει μία σειρά από παρεκκλήσει, Για παράδειγμα, ε, τη σήμερον ημέρα, εάν ε, το αλίευμα είναι χαμηλότερο από 50 κιλά, το σκάφος δεν υποχρεούται να το αναφέρει. Ε, δεν ισχύει πλέον λοιπόν αυτή η εξαίρεση, αυτή η παρεκκλήση. Δηλαδή όλα τα σκάφη τα πρέπει να κάνουν τη σχετική αναφορά, συμπεριλαμβανομένου και του μικρού μεγέθου, των μικρών, μικρού μεγέθους ε, σκαφών. Επίσης, υπάρχει ε, και η εξαίρεση ό,τι αφορά τις ε, πωλήσει ε, για μη καταχωρημένους, μη εγγεγραμμένους αγοραστούς και υπάρχει μια προσαρμογή των κανόνων σε ό,τι αφορά τις ανοχές ανάμεσα δηλαδή στα προβλεπόμενα δεδομένα αλλιευμάτων και στις πραγματικά εκφορτώμενες ποσότητες. Αλλά δεν θα μπω τώρα στις τεχνικές λεπτομέρειες. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του συστήματος ζήγησης, στάθμισης δηλαδή των αλλιευμάτων, ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι, πόροι τελικά, οι θαλάσσιοι πόροι οι οποίοι έχουν εξαχθεί από τη θάλασσα. Ε, βλέπουμε πως το σύστημα το σημερινό, οι σημερινές διατάξεις δεν ανταποκρίνεται στις, στις ανάγκες μας. Οπότε λοιπόν προτείνουμε όλα τα αλλιέματα, όλα τα προϊόντα αλλιές να ζυγίζονται κατά την εκφόρτωσή τους. Ε, ανεξαρτήτως του ποιο είναι ο οικονομικός φορέας ο οποίος είναι κατοχωρημένος στο κράτος μέλος, δηλαδή αν είναι ο ίδιος αλλιές ή κάποιος άλλος. Επίσης έχουμε Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά την ε, αναφορά των παρεμπίπτων των αλλιευμάτων, προσπαθούμε να είμαστε πιο ακριβείς και επίσης να ορίζουμε τις ευθύνε ε, των διαφόρων οικονομικών φορέων ακριβώς σε ό,τι αφορά τη ζήγηση τόσο έπλο όσο ε, και στην ξηρά. Ένα τρίτο κομμάτι τώρα αφορά αυτό που είπαμε, την γεβήρωση του χάσματος με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Καταρχήν εδώ έχουμε να κάνουμε το ζήτημα ε, των ε, υποχρεώσεων εκφόρτωση. Δηλαδή παρότι ισχύει η υποχρέωση εκφόρτωσης σήμερα ημέρα, δεν υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες ω προς το πώ ακριβώ γίνεται ο έλεγχο τη υποχρέωση εκφόρτωση. Εδώ λοιπόν εμεί προτείνουμε την υποχρεωτική χρήση CCTV, δηλαδή τηλεόραση κλειστού κυκλώματο, σε ό,τι αφορά τα επιμέρους σκάφη και κομμάτια ε, στόλων, τμήματα στόλων, με βάση ακριβώ το επίπεδο κινδύνου και η εφαρμογή αυτή θα γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο στα, κράτη-μέλη, συγγνώμη, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ίσου κανόνε του παιχνιδιού για όλου. Επίση, προτείνουμε μια σειρά από βελτιώσει στο σύστημα ελέγχου ε, της ικανότητα. ικανότητας. Δηλαδή, ε, ε, σήμερα στον κανονισμό ελέγχων ε, προβλέπονται μια σειρά από διατάξει, οι οποίε όμω δεν είναι αποτελεσματικέ και ούτε εφαρμόζονται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Εδώ λοιπόν εμεί προτείνουμε την απλούστευση του συστήματο για τον έλεγχο ε, της αλλιευτικής μέσω συνεχούς παρακολούθησης ε, και ελέγχου ε, της ισχύω ε, του κινητήρα με βάση τα είδη των αλευτικών σκαφών. Επίσης προτείνουμε μια, ακολουθούμε μια σειρά από που έκανε το ελεκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την επαλήθευση ακριβώς ε, του, της ισχύω των κινητήρων. Από εκεί και μετά ένα ε, τέταρτο κομμάτι είναι οι συνέργειες με άλλους ε, τομείς πολιτικής και ειδικότερα δε, τον, την πολιτική προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ λοιπόν προβλέπουμε υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την αναφορά των αλληλευτικών εργαλείων, τα, οι οποίες απώλειες θα αναφέρονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού δηλαδή ημερολογίου σκάφους. τη σήμερα ημέρα αυτό δεν γίνεται ηλεκτρονικά γίνεται στο ημερολόγιο, δηλαδή σε έντιμη μορφή και συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν γίνεται καν η αναφορά για τα απολεσθέντα αυτά εργαλεία ε, σε μια σειρά από κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν με αυτή τη νέα διάταξη ελπίζουμε πως θα είναι πιο εύκολη η αναφορά. Επίσης προτείνουμε ένα νέο και πολύ πιο διευρυμένο ορισμό ε, των ε, παγωμένων περιοχών, των restricted area, ε, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών σε επίπεδο κράτους μέλους ή και σε ευρύτερο επίπεδο και οι νέοι κανόνες σε ό,τι αφορά ακριβώς την παρακολούθηση των αλληλευτικών σκαφών σε κάθε περίπτωση θα βελτιώσουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλληλευτικών σκαφών στι απαγορευμένε περιοχέ. Πράγμα που τη σήμερα ημέρα είναι δύσκολο γιατί ακριβώ δεν μπορούμε να παρακολουθούμε, να ανενεύουμε δηλαδή αυτά τα αλευτικά σκάφη και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν δραστηριοποιούνται ή όχι μέσα σε μια απαγορευμένη περιοχή. Ένα ε, ακόμα κομμάτι της συνέργειας είναι η συνέργεια με την πολιτική στον τομέα ε, της, ε, της πολιτικής για την ασφάλεια των τροφίμων. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε καλύτερη ειχνασιμότητα των τροφίμων ειδικότερα σε ό,τι αφορά την μεγαλύτερη συσχέτιση ανάμεσα σε κάθε αλευτικό ταξίδι αφενό και ε, τα, τις εκφορτώσεις, τα λιεύματα δηλαδή, σε σχέση με αυτό το ταξίδι αφετέρου και προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τις νέες διατάξεις και στα εισαγόμενα είδη αλλά και σε όλα τα, ε, τα, τα αλλιεύματα αλλά και τα οστρακοειδή τα οποία έχουν τύχει περαιτέρω επεξεργασίας. Και επίσης προσπαθούμε και εδώ να εισαγάγουμε κανόνες σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση των σχετικών δεδομένων και για κατάργηση ε, όλων των πληροφοριών σε έντυπη μορφή σε αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν τις τροποποιήσεις που θα λάβουν χώρα σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τους ελέγχους. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τον ε, κανονισμό για την ε, ίδρυση της ΕΦΚΑ, ουσιαστικά διατάξεις στοχεύουν την πλήρη ευθυγράμμιση των στόχων και της αποστολής της ΕΦΚΑ στην κοινή αλληλευτική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και τη εξωτερική διάσταση αυτής της πολιτικής. Επίσης ε, προσπαθούμε να διευρύνουμε το ε, γεωγραφικό ε, πεδίο αναφοράς, αν θέλετε, της εντολής της αρχής, γιατί τη σήμερα ημέρα είχε να κάνει μόνο με διεθνή ύδατα και όχι με ευρωπαϊκά ύδατα. Τώρα θα ισχύει και για τα ευρωπαϊκά ύδατα. Και επίσης προσπαθούμε να έχουμε περισσότερες δυνατότητες λήψης αποφάσεων για τον ΕΦΚΑ σε ό,τι αφορά και περαιτέρω συμφωνίες και ε, με περαιτέρω επιδοτήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, κανονισμό για την αλληλεία IUU, προσπαθούμε να ε, ψηφοποιήσουμε το πιστοποιητικό αλληλεία, το CATS όπω λέγεται. Και προσπαθούμε λοιπόν σιγά σιγά να περάσουμε στην ψηφιοποίηση αυτού του εντύπου CATS. Έτσι λοιπόν αυτό ο νέο κανονισμό θα δώσει τη νομική βάση για να περάσουμε στην ψηφιακή μορφή του ΚΑΤΣ. Και επίση οι διατάξει όπω είπαμε οι οποίε περιλαμβάνονται σήμερα στον κανονισμό IUU και αφορούν κυρώσει θα περάσουν μελλοντικά, θα συμπεριληφθούν μελλοντικά στον κανονισμό για του ελέγχου. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια και σε ό,τι αφορά την ημερομηνία θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού ε, που προτείνεται από την Επιτροπή. Εμείς λοιπόν προτείνουμε οι ε, αλλαγές που θα αφορούν τον κανονισμό για την ίδρυση ε, του ΕΦΚΑ να τεθούν σε ισχύ άμεσα. Σε ό,τι αφορά όλε τι υπόλοιπε τροποποιήσει, δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να γίνει η προσαρμογή τη δευτερογενού ε, νομοθεσία. Δηλαδή σε ό,τι αφορά τι κατεξοδότητε αλλά και τι εφαρμοστικέ πράξει. Και επίση δίνουμε αυτή την ε, διάμεση περίοδο ώστε να υπάρξει η ε, δημιουργία, η ανάπτυξη των σχετικών ψηφιακών εργαλείων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα αλληλευτικά σκάφη μικρού μεγέθου. Και γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε ω έναρξη ισχύω 24 μήνε μετά την έγκριση του κανονισμού. Όλοι νομίζω πως γνωρίζετε τώρα τη διαδικασία της συναπόφησης, όπως αναφέρθηκε δηλαδή ήδη από τον πρόεδρο, αναφέρθηκε ήδη ότι θα πρέπει να γίνει δηλαδή εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το Συμβούλιο από τη δική του πλευρά εξετάζει στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την εσωτερική και εξωτερική αλληλεία αυτό το ζήτημα και το μόνο θέμα που παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα είναι οι κυρώσει και οι παραβάσει. Ε, στον ιστότοπό μα εδώ σε αυτήν την ιστοσελίδα βλέπετε όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε φορτώσει που εξηγούν ακριβώ τη συλλογιστική πίσω από τι προτάσει, ε, την αξιολόγηση αντικτύπου, τη διαβούλευση που έλαβε χώρα, την έκθεση που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα λοιπά. Αυτή λοιπόν είναι η ιστοσελίδα. Αυτά από την πλευρά μου. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Αγγιλέρα είπε ότι θα είναι συγγήτρια, έτσι δεν είναι. Και θα δώσω και στον κύριο τη το λόγο για ερωτήσει, αλλά έχω και εγώ μια ερώτηση πρώτα απ' όλα, που έχει να κάνει με την πρόταση για το ελάχιστο επίπεδο προστήμων. Αναγκαία πρόταση, αλλά το Συμβούλιο, φαντάζομαι, θα θεωρεί ότι παρεμβαίνεται στην εθνική δικαστική ανεξαρτησία ή ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ερώτηση. Λοιπόν, στη συζητήσεις στο Συμβούλιο Ακόμα είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο. Εξετάζουμε άρθρο-άρθρο τον κανονισμό. Οπότε δεν υπάρχει ακόμα θέση, τοποθέτηση στο Σεβούλιο που θα μπορούσε ε, να έχει νόημα. Πρέπει να είσαστε υπομονετικός, ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Αλλά αυτό που ακούμε από τις χώρες μέλη, δεξιά και αριστερά, είναι ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε σε θέματα τα οποία θεωρούνται ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας. Μα δεν είναι αυτή η, πρόταση, η πρόθεση της πρότασης. Η πρόθεση της πρότασης είναι να υπάρχουν διοικητικές διαδικασίες στα σύνορα και επιπλέον οι χώρες μέλη, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να εφαρμόσουν ποινικέ διατάξεις σύμφωνα με τους δικούς τους κανονισμούς προεδροσμό. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή κατά το παρελθόν είχε κάνει προτάσεις σε σχέση με την θέση σε εφαρμογή τέτοιων διατάξεων. Αλλά όταν φτάνουμε στα εθνικά δικαστήρια, εκεί τα πρόστιμα ε, διαφέρουν πάρα πολύ. Καταλαβαίνω, θέλω να πω, τη δυσκολία που έχετε για την εφαρμογή τέτοιων προτάσεων. Κυρία, ο κύριος Ματίτς. Παρακαλώ κύριε Ματίτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μιλάω εκ μέρους τη συναδέρφου Κλάρα Ντουλέρα. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσει την συνάδελφο Ιζαμπέλ Τομάς από τη Σοσιαλιστική Ομάδια που κατά την προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφοσιώθηκε σε αυτό το φάκελο. όπω όλοι γνωρίζετε, σοφά αποφάσισε να σταματήσει η διαδικασία του φακέλου αυτού, προκειμένου να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα στη θέση της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το σημαντικό θέμα. Η Κλάρα δέχεται λοιπόν την πρόκληση να είναι η συγγήτρια για αυτή τη σημαντική υπόθεση και εκφράζει την επιθυμία ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε συνένεση ώστε να καταλήξουμε σε μια ισχυρή θέση μας απέναντι στα άλλα ε, θεσμικά όργανα. Από αυτού λοιπόν η διαδικασία πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή. Με άλλα λόγια θα συντάξει νέα έκθεση που θα παρουσιαστεί στην ε, Επιτροπή και θα υπάρξει φυσικά και ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. Η κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να αποφασίσει να επανακαταθέσει τις τροπολογίες που έχει ήδη καταθέσει ή να προτείνει νέες τροποποίησεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κανονισμό. Οι προθεσμίες δεν έχουν τεθεί ακόμα, αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει το χρόνο που τους χρειάζεται ώστε να προβεί σε διαβουλεύσεις και να παρακολουθήσει όλες τις συζητήσεις προκειμένου να εκπονήσει την τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ζητά συγγνώμη που δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά της είναι αδύνατο να παρακολουθήσει ταυτόχρονα δύο συνεδριάσεις. Είναι στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας. Όπως ξέρετε, δημόσια ακρόαση θα υπάρξει για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Ελίας τον Οκτώβριο. Και επί τη ευκαιρία αυτή θα έχουμε χρόνο για συζήτηση. Οπότε η Κλάρα δεν θέλει τώρα να περάσει σε λεπτομέρειες. Αυτό που θα ήθελε όμως είναι να πει ότι πιστεύει πως είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η πρόταση και να συμπληρωθεί βάσει του στόχου που είναι η απλοποίηση, να το κάνει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη θα ήθελε να υπογραμμίσει και την αναγκαία αναρμόνιση προκειμένου να μην δημιουργηθεί η αίσθηση αδικίας απέναντι στους αλλοί των διαφορών χωρών. Επιπλέον πρέπει να στηρίξουμε και τη δημιουργία ενός μηχανισμού οικονομικού αλλά και ελέγχου και να προβλεφθούν και διατέξεις που θα αντικατοπτρίσουν τις ανάγκες και τις ε, υδατοκαλλιέργειας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση που είναι να ενισχύσουμε το σύστημα ελέγχων και επιθεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς από την άλλη μεριά να αυξηθεί το διοικητικό άχθος και οι προσπάθειες που κάνουν οι χώρε μέλη. Κλάρα πιστεύει ότι ο εξυγχρονισμό και η χρήση νέων τεχνολογιών πρέπει να οδηγήσουν στην ε, υποχρέωση ε, αναφοράς των εκφορτώσεων πάντα, αλλά και την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της υπηρεσίας της ίδιας ελέγχου ε, αλίας. Αλλά αυτό να γίνεται και με τρίτες χώρες σε όλους τους τομείς της αλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Μιλμάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινάμε με τον έλεγχο, που είναι ένας πολύ σημαντικός φάκελος. Έλαβα γνώση και στην προηγούμενη θητεία, γιατί ήμουν ασκιώδης εισηγητής και ασχολήθηκα με αυτόν. Ξέρω ότι ο κανονισμός είναι πολύ σημαντικός και θέλω να ευχαριστήσει την Ιζαμπέλ Τόμα που ήταν η εισηγήτρια στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σίγουρα όταν η Κλάρα Αγγιλέρα μας φέρει την έκθεσή της θα καταλάβουμε περισσότερο. Τώρα όμως έχω να κάνω μερικά σχόλια, χωρίς να θέλω όμως να μακρηγορήσω πολύ, γιατί προτιμώ να ακούω την Επιτροπή και να την ευχαριστήσω επ' ευκαιρία που μας παρουσίασε και πάλι την πρότασή της. Το κείμενο μου φαίνεται περίπλοκο, χρειάζεται να το μελετήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω επίσης, όπως και η Κλάρα, ότι είναι καλό να υπάρχει ομοιογένεια στο καθεστώς κυρώσεων. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Γιατί είμαστε σε μια κατάσταση ανισορροπίας. Ο κανονισμός αποτελεί περισσότερο μια οδηγία που δεν έχει ενσωματωθεί ως ε, τέτοια στη νομοθεσία των χωρών μελών. Υπάρχουν δηλαδή τεράστιες διαφορές όταν εφαρμόζονται κυρώσεις μεταξύ των χωρών και λειτουργεί περισσότερο σαν οδηγία, όπως είπα και πριν, και όχι ως κανονισμός. Γι' αυτό, τον υπάρχει ένας ε, νέος κανονισμός που να είναι πραγματικά κανονισμός και νομιογενή όλο αυτό το θέμα, το τόσο λεπτό του ελέγχου και των κυρώσεων, είναι σημαντικό και επίσης ξαναφτιάχνεται λίγο έτσι και ε, ομιγενοποιείται. Φυσικά και θα πρέπει προσεκτικά να μελετήσουμε την πρόταση αυτή, αλλά πάντως ο κανονισμός σε θέματα ελέγχου με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών κλπ. δεν θα πρέπει να αποτελεί γραφειοκρατικό και οικονομικό περί το βάρος. Πιο πολύ αυτό απασχολεί την μικρή ε, κλίμακας ε, αλία. Όλες αυτές οι καινοτομίες, τεχνολογία κτλ. Ε, δεν είναι κάτι που ακούνε με ενθουσιασμό οι αλλιείς μικρής κλίμακας, αλλά μάλλον με επιφυλάξεις και δισταγμούς. Έπειτα υπάρχει και το θέμα του κόστους. Και υπάρχει και το θέμα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί με τον κύριο Ματσάδο, δηλαδή το θέμα των ε, κλειστών κυκλωμάτων ε, τηλεόρασης, που και αυτό είναι πολεμικό ζήτημα το κατά πόσο σε ένα ιδιωτικό χώρο τελικά υπάρχει δίσδυση απ' έξω. Είναι ένας χώρος όπου ζει επίσης κανείς, δεν εργάζεται μόνο. Τίθεται και το θέμα της ε, χρησιμότητας τέτοιων ε, ε, εξοπλισμών κλειστού κυκλήματος. Μήπως είναι υπερβολικά δυσδυτικό δηλαδή αυτό το σύστημα. Όταν έρθει η ώρα να διαλέξουμε, ίσως πρέπει να δούμε με τον κίνδυνο. Αυτά που είναι πάνω από 18 μέτρα, εκεί ελοχεύει μεγαλύτερος κίνδυνος. Ε, θεωρούνται ένοχα αυτά τα σκάφη εκ προημίου. Είναι λεπτό το ζήτημα. Έπειτα υπάρχει και η θέληση να μετράμε συνέχεια την, ε, τις δυνατότητες που έχει ένα σκάφος όταν υπάρχουν ε, ποσοστώσεις υπάρχουν όποιε και αν είναι οι δυνατότητε των σκαφών. Οπότε το θέμα δεν έχει να κάνει τόσο με την ελεία όσο με την ασφάλεια. Και κάτι ακόμα, γιατί όπως είπα δεν θέλω να μακρηγορήσω, πρέπει να υπάρχει έλεγχος και της αλίας για ψυχαγωγία. Θα είναι δύσκολο βέβαια, γιατί πρόκειται για τεράστιο όγκο και πώς θα ελεγχθεί αυτός ο όγκος. Αλλά είναι καλό στον τομέα αυτό που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και ποσοτικά να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος. Και αυτά τα πιστοποιητικά επίσης αλλιεύσει πιστεύω ότι είναι σημαντικά για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα ε, τις εισαγωγές που έχουμε από τρίτες χώρες. Έτσι θα υπάρχει μια ισορροπία και ό,τι έρχεται απ' έξω να μην ε, χρησιμοποιείται σαν ε, κόλπο για να καλύπτονται παράνομα αλλιεύματα. Θα δώσουμε μεγάλη σημασία λοιπόν σε αυτήν την νέα πρόταση και θα υποβάλουμε ό,τι τροπολογίες κρίνουμε ε, καλό. Αποφασίσαμε για μια ακρόαση, δημόσια ακρόαση για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα την κάνουμε τον Οκτώβριο και πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό αυτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Η πρόταση προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχουμε στο πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικό έλεγχο της αλλιευτικής δραστηριότητας και την βιώσιμη διαχείριση των πόρων. Προσπαθούμε επίσης να απλωστεύσουμε και να βελτιώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο των ελέγχων. Η πρόταση κανονισμού δείχνει όμως να αγνοεί τι ιδιαιτερότητες τη μεσογειακής αλίας, με στόλο από μικρά σκάφη κυρίως, και επομένω οι κανόνε ελέγχου πολύ δύσκολο θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά στην πραγματικότητα. Μεταξύ αυτών, για παράδειγμα, ε, μιλώ για τις υποχρεωτικές ε, κάμερες CCTM, για τις υποχρεωτικές εκφορτώσεις. Αυτό θα ήταν ε, ένα σημαντικό άχθος για τις επιχειρήσεις και θα ήταν μέτρα αποτελεσματικά, οικονομικά μη παραγωγικά και κυρίως μη υλοποιήσιμα ιδιαίτερα και επαναλαμβάνω για τις ιδιαιτερότητες της μεσογειακής Αλληλεία. Επίση, υπάρχει μια διαφορά με το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων και τη ιδιωτικότητά του. Επίσης μιλούμε για τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μητρώου και ένα σύστημα γεωεντοπισμού για τα σκάφη, για τη διαχείριση, αλλά το EMFF δεν προβλέπει χρηματοδότηση σχετικά κονδύλια ε, ε, για κάτι τέτοιο, όπως μας είπε και ο Γενικός Διευθυντής Ματσάδο νωρίτερα. Επίσης φαίνεται να έχουμε τεχνικές ε, ιδιαιτερότητες που πολύ δύσκολα μπορούν να βρουν ομοιόμορφη υλοποίηση, διότι τα υποκείμενα είναι τελείως διαφορετικά. Για παράδειγμα, να είναι ανάλογη η κύρωση προς την οποιαδήποτε παράβαση ε, τη στιγμή μάλιστα του, του εντοπισμού της παράβασης. Δεν υπάρχει σαφήνεια ε, νομοθετική και δεν υπάρχει ομοιόμορφη και δίκαιη ε, εκτέλεση, υλοποίηση αυτών των, του συστήματος αυτού κυρώσεων. Ελπίζω, εν πάση σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε μια αποτελεσματική συνεργασία με τους συναδέλφους της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you. Mrs. Ε, ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα μιλήσω γαλλικά. Δύο ερωτήσει έχω. Περιμένοντα να ξαναρχίσει η διαδικασία αναθεώρηση ε, του κανονισμού για τον ελέγχο, θέλουμε να υπογραμμίσουμε κάποιε πτυχέ που πιστεύουμε ότι πρέπει να προσέχουμε συνεχώ. Η διαφάνεια πρέπει να αποτελεί στοιχείο κλειδί του μελλοντικού κανονισμού όσον αφορά τον ελέγχο τη Αλλία. Να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου και για τι κυρώσει που επιβάλλονται και για του λόγου για του οποίου επιβάλλονται ε, η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να δημοσιεύει τις εκθέσεις της ελέγχου για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν τον κανονισμό οι χώρες μέλη συμπεριλαμβανομένου και του κανονισμού ελέγχου. Έπειτα, ενώ ισχύει εδώ και 10 χρόνια ο κανονισμό για τους ελέγχους, ελάχιστες χώρες έχουν εφαρμόσει πραγματικά αποτρεπτικέ κυρώσει. Ο αριθμό των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί είναι πολύ χαμηλό. και το επίπεδό του δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που αναφέρονται στον ε, κανονισμό. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε σε μια εκθεσή της ότι τα μέτρα εφαρμογή κυρίως όσον αφορά τις κυρώσεις και το σύστημα πόντων μετά από παραβάσεις ε, είναι γεμάτες ε, ελλείψεις. Οι χώρες μέλη λοιπόν θα πρέπει να πιεστούν να εφαρμόσουν τον κανονισμό ελέγχου και τον ΙΕΝΕΝ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει δράση για να καταλάβει γιατί γίνονται όλα αυτά και να τα διορθώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, αυτή είναι η ερώτησή μου. Πώς θα βελτιώσει αυτή την κατάσταση στο μέλλον και μέτρα ισχυρά κατά των χωρών μελών, όπως για παράδειγμα ε, κατά παραβάση προβλέπει να τα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε. Όλοι συμφωνούμε ότι η έκθεση αυτή θα είναι αρκετά περίπλοκη. Ήταν ήδη περίπλοκη στην προηγούμενη θητεία, θα είναι και εδώ. Ελπίζω να τα καταφέρουμε καλύτερα αυτή τη φορά. Πάντως, βάσει των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί και το ένα είναι τα δεδομένα που έχουμε από την Αλία που δεν είναι επαρκή, είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται και διαφορετικές κυρώσεις αν εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τι βαθμό έχουμε δεδομένα ή τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των χωρών μελών για να εντοπίσουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Γιατί σίγουρα κάποιες χώρες θα έχουν κάνει προσπάθεια παραπάνω για να ε, καλύψουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, άλλες πολύ λιγότερο. Οπότε τελικά ε, φτάνουμε στο περίπου να ποινικοποιούμε τον ελληνικό κλάδο, κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Γι' αυτό και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια ώστε να εντοπίζουμε σωστά τα προβλήματα και έτσι να υιοθετούμε και τα κατάλληλα μέτρα. Κατόπιν τούτο, συμφωνώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη συλλογή δεδομένων και τα δεδομένα μας. Πρέπει να βοηθήσει σε αυτό ο ίδιος ο κλάδος. Έπειτα έχουμε εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κλάδος θέλει να ζήσει από τη θάλασσα και από την αλία ζει. Οπότε ο κλάδος ο ίδιος έχει κάθε συμφέρον να υπάρχουν οι κατάλληλοι έλεγχοι. Οπότε μπορούμε να βασιστούμε σε αυτούς, πιστεύω. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε. Έχοντας υπόψη μας τα σχέδια διαχείρισης που εγκρίναμε στην προηγούμενη θητεία και τις δυσκολίες που είχαμε μερικά από αυτά, θέλω να ξέρω, η διαφορά απαιτήσεων συγκρίνοντας τα σχέδια δεν στρεβλώνει την κατάσταση. Τελικά θα έχουμε έναν κανονισμό που θέλουμε να ισχύει εξίσου παντού. Κι όμως στη Βαλτική οι επιπτώσεις ήταν μάλλον αρνητικές. Τώρα για την ψυχολογική αλία, ναι, συμφωνούμε ότι πρέπει να ελέγχεται και αυτή. Αυτό το καυγά τον είχαμε στην προηγούμενη θητεία. Και για την υποχρέωση δήλωση εκφορτώσεων. Διαβάζουμε τελευταία επιστημονικές εκθέσεις που θέτουν υποαμφισβήτηση το σύστημα των εκφορτώσεων αυτών. Εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να πετύχουμε ένα στόχο. Γι' αυτό υπήρξε και μείωση ποσοστώσεων όσον αφορά την αλίευση από διάφορα σκάφη, αλλά και κυρίως γιατί δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε αρκετά την αλία. Γι' αυτό θέλω να ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλύσει τις εκθέσεις αυτές, ε, προβληματίζονται, πιστεύουν ότι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε κάτι παραπάνω σε αυτόν τον κανονισμό ελέγχου. Και τέλος, για το θέμα της εχνηλασιμότητας. Συμφωνούμε απόλυτα και ζητάμε να γνωρίζουμε τι γίνεται με κάθε ψάρι από τη στιγμή που βγαίνει από τη θάλασσα μέχρι που φτάνει στην κονσέρβα. Γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για τρόφιμα, πρόκειται για δικαιώματα ε, των καταναλωτών. Μερικές φορές δεν γνωρίζουμε ε, κάποιες κονσέρβες από που προέρχονται. Και γι' αυτό και θέλουμε ρύθμιση για να προστατεύσουμε τον κλάδο μικρής κλίμακας αλίας ή τους πιο αδύναμους αλής. Μπορεί να υπάρχει προϊόν ποιότητας, αλλά όταν φτάνει στον καταναλωτή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει αν το προϊόν που έχει αγοράσει έχει αλλιευθεί με, ε, κλίμακα, με μικρής κλίμακας αλεία ή έχει αλλιευθεί με βιομηχανική αλεία. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να υπάρχει υποχρέωση ετικέτας και στις κονσέρβες. Αυτό θα βοηθήσει την αλία μικρής κλίμακας να αξιοποιήσει καλύτερα την παραγωγή της χωρίς να ανταγωνίζεται με άλλα προϊόντα που δεν λέω ότι είναι κακά. Καλά είναι, οι κονσέρβες είναι μια χαρά. Αλλά εγώ που είμαι καταναλωτής θα ήθελα να γνωρίζω όταν πληρώνω τι αγοράζω ακριβώς. Μία έκθεση που έγινε πριν από τρία χρόνια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι υπάρχουν απάτες πολλές φορές με τις κονσέρβες γιατί δεν ξέρουμε τελικά τι αγοράζουμε ακριβώς. Γι' αυτό ρωτάω, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε και σε αυτό. Εγώ πιστεύω πως θα έπρεπε. Και εννοείται ότι θα συνεργαστούμε όλοι για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά είναι αναγκαίο, νομίζω, να βασιστούμε περισσότερο στον ίδιο τον αλληλευτικό κλάδο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστούμε. Δεν έχω άλλους ομιλητές. Mr. Miramon, you wanted to speak on behalf of uh, Mr. von Dalen? Eso es, gracias. Es que... Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο κύριος Βαντάλεν δεν μπορούσε να είναι εδώ για λόγω δυσάριστων προσωπικών ε, ε, λόγων. Ε, μου ζήτησε λοιπόν να διαβιβάσω τη θέση τη δική του και της Ελλανδικής Αντιπροσωπείας. Ε, αναφέρομαι στον κανονισμό ελέγχου και μεταφράζω. Ε, λέγει ότι η φυστάμενη πρόταση είναι εκτός του πλαισίου που είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει. Πρέπει να έχουμε ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο. Για την Ολλανδία ο όγκος των εφορτώσεων είναι πολύ σημαντικό και έχουμε εξαιρέσει σήμερα που επιτρέπει στου αλληλείς να αλλιεύουν ει το σκάφο τα αλλιεύματα. Και αυτό γίνεται αν έχουμε εξοπλισμό πιστοποιημένο που είναι μια καλή λύση για την Ολλανδία διότι το βάρος είναι πολύ διαφοροποιημένο Η ζήγηση λοιπόν επί του σκάφους είναι πολύ διαφοροποιημένη ανάλογα με τον εξοπλισμό από χώρα σε χώρα. Ο, ο, ο εξοπλισμός που απαιτείται λοιπόν είναι σημαντικός αναλόγως μάλιστα με το λιμάνι στο οποίο εκφορτώνει. Θα ήθελε η Ολλανδική Αντιπροσωπεία λοιπόν να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το συγκεκριμένο αυτό πρόβλημα και προσθέτει ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε μια εναρμόνιση σε, ως προς τις κυρώσεις. Οι Ολλανδοί είναι πολύ αυστηροί σχετικά με την αποτελεσματική υλοποίηση των ελέγχων, αλλά πολύ συχνά οι αλληλείς ακούν φήμες ότι σε άλλες χώρες δεν γίνεται το ίδιο. Και επομένως τους διαβιβάζεται μια αίσθηση αδικίας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εναρμόνιση των κυρώσεων για να έχουμε πιο αποτελεσματική υλοποίηση της νομοθεσία των ελέγχων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ναι, ε, δεν σας είδα, παρακαλώ. Έχετε το λόγο, ε, ε, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να αναφερθώ στο σχεδίο διαχείρισης της Βαλτικής και πάλι καλά που έχουμε εδώ τους αρμοδίους. Όχι, στην Αδριατική αναφέρομαι. Ε, ζητώ συγγνώμη, λέει η ομιλήτρια. Στην Αδριατική αναφέρομαι. Αναφέρθηκα νωρίτερα, δηλαδή διορθώνω. Ε, προτού απαντήσει η Κομισιόν, λέει ο Πρόεδρο, να προσθέσω και εγώ ένα-δύο στοιχεία. Για τι κάμερε, τα τηλεοπτικά στήματα. Νομίζω ότι ο Σκοτσέζικο στόχο είχε εξοπλιστεί πριν από κάποια χρόνια με κάμερε και έλαβε μια ενισχυμένη ποσόστοση ω αντιστάθμιση. Επομένω, υπάρχουν διάφορα συνδεδεμένα ζητήματα και ρωτώ, η σχετική μελέτη που είχε γίνει τότε μπορούμε να την έχουμε. Εγώ δεν την είχα δει. Επίσης για την επιβολή εκθέσεων για εξοπλισμό που έχει απολεστεί, για αλλιευτικό εξοπλισμό. Αυτό πώς το αντισταθμίζεται, πώς το αποζημιώνετε; και τι κυρώσεις αναλαμβάνεται για σκάφη που χάνουν τον αλλιευτικό του εξοπλισμό, τα αλλιευτικά της μέσα. Υπάρχουν κυρώσεις σχετικά με αυτό. Και αν δεν υπάρχουν, και, και μάλλον αν υπάρχουν κυρώσει, γιατί δεν έχουν αναφερθεί, γιατί δεν τις ε, γνωρίζουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τα κρατημέλη για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Τις έχουμε σημειώσει προσεκτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να πάμε σε λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τις διάφορες πτυχές που υπευλήθησαν πράγματι υπάρχει μια αίσθηση ότι το σύστημα του ελέγχου και των κυρώσεων πρέπει να είναι εναρμονισμένο ώστε να είναι ισότιμο το παιχνίδι. Και αυτό είναι από τι βασικότερε εστιάσεις μα, ότι δηλαδή οι αλληλείς θα λαμβάνουν ίση μεταχείριση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Άκουσα κάποιε ανησυχίε. για αυξημένο διοικητικό άκθο ή εν για μεγαλύτερο άκθος για τους επιμέρους αλείς. Αυτή δεν είναι καθόλου η πρόθεσή μας. Ιδιαίτερα για τους μικρής κλίμακα τόλους, δεν προτείνουμε να αποτυπωθεί το ίδιο επίπεδο λεπτομέρειες που επιβάλλουμε για τους μεγαλύτερους τόλους. Για τους μικρούς τόλους προτείνουμε εύκολα και φθηνά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι αλείς ώστε να καταγορήσουν τα δεδομένα αλίευσής τους. Από τις εκθέσεις μας γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε υποχρεώσεις εντύπων λόγω της διαρκούς επανασυμπλήρωσης και επανασυμπλήρωση των, εντύπων έχουμε εξαιρετική πρακτική διοικητική καθυστέρηση και κόστο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο θα ανεβάζει απευθεία τα δεδομένα αυτά στο κεντρικό σύστημα το οποίο σίγουρα θα είναι λιγότερο επαχθές. έχω και άλλα παραδείγματα για να σας πείσω ότι καθόλου δεν είναι η πρόθεσή μας να έχουμε μεγαλύτερο κόστος στους αλληλείς των διαφόρων χωρών. Για την ποινικοποίηση που αναφέρθηκε. Επίσης καθόλου δεν είναι η πρόθεσή μα. Τι είναι αυτό που λέμε. Μιλούμε για τη χρήση από πλευρά των αλλιέων μιας κοινή πηγής πόρων και δεδομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιείται με υπεύθυνο τρόπο από όλους τους αλληλείς Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι όλοι θα σε μορφούνται προς τους κανόνες και θα εμπιστεύονται τους συναδέλφους τους. Για τις κάμερες ε, των κλειστών κυκλωμάτων δεν μιλούμε καθόλου για ποινικοποίηση. Δεν είναι αυτή η πρόθεση. Είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρούνται οι κανόνες. Ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Ματσάδα, το είπε το πρωί. Δεν πρόκειται να εισβάλλουμε στην ιδιωτικότητα των αλλιέων. Θα εξασφαλίζουμε ότι οι κάμερες σαρώνουν μόνο τα σημεία του σκάφους που λαμβάνει χώρα η αλευτική δραστηριότητα, όχι τα εσωτερικά, όχι τις καμπίνες του προσωπικού, του πληρώματος. Μόνο για τις χρήσεις των ελέγχων και των επιθεωρήσεων. Με χαρά να συζητήσουμε ενδελεχέστερα, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια μαζί σας για τα θέματα αυτά και για την ερώτησή σας, Πρόεδρο, για τη χρήση των καμερών αυτών CCTV είχαμε κάποια πιλωτικά σε συγκεκριμένες αλευτικές ζώνες και στα πιλωτικά αυτά προγράμματα αποφάσισαν τα κρατη να δώσουν κίνητρο. Έχουμε τα αποτελέσματά τους και μπορούμε να δούμε κατά πόσον έχουμε ένα, έγγραφο σύνοψης που θα μπορούσαμε να στο διαθέσουμε για τα πορίσματα αυτά. Αυτό που προκύπτει με σαφήνεια είναι ότι το CCTV είναι αποτελεσματικό για τον έλεγχο των υποχρεώσεων εκφόρτωσης. Και είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο έχουμε εξετάσει. Ήθελα επίσης να αναφέρω το εξής. Μας ρωτάτε ποιος θα αναλάβει το κόστος. Υπό το παρόν e MFF έχουμε 680 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν μόνο στην χρηματοδότηση εργαλείων ελέγχου που είναι διαθέσιμη για τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των επιχειρησιακών και υπό την παρούσα χρηματοδοτική περίοδο. Για το μέλλον, είχαμε προτείνει ότι πολύ σημαντικό τμήμα του e MFF μπορεί να χρησιμοποιείται για χρήση ελέγχου, περίπου το ίδιο ποσό, και για το μελλοντικό EMFF είχαμε πει ότι για τις μικρές κλίμακες θα πρέπει να έχουμε χαμηλότερη ποσόστοση για τις συσκευές αυτές τις τηλεοπτικές, τις κάμερες. Έχουμε προβλέψεις λοιπόν υπό τα, υπό τα χρηματοδοτικά μέσα. Τώρα πρόεδρε, είναι δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς ότι η υποβολή εκθέσεων θα, γίνεται σεβαστή σε κάθε περίπτωση, ειδικά σε πρώτο χρόνο ε, ενημέρωσης για τις κυρώσεις του περσινού έτους μπορώ να σας πω ότι όλοι αυτοί που απόλυσαν αλλιευτικά μέσα δεν τα απόλυσαν επίτηδες. Είχαμε φρουτούνες στη θάλασσα, τρικυμίες και τα λοιπά, ατυχήματα. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως. Έγινε και άλλη μια ερώτηση, αν σημείωσα σωστά. Τι κάνουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη υλοποιούν το σύστημα ελέγχου αποτελεσματικά Εμείς προχωρούμε σε συστηματικές ε, εκθέσεις ελέγχου, ελεγκτικές, για να εξασφαλίζουμε ότι τα δικά του συστήματα ελέγχου συμμορφούνται προς τους κανόνες. Και όταν έχουμε οποιαδήποτε ένδειξη στην έκθεση, αναλαμβάνουμε την δράση που απαιτείται. Μπορεί αυτή να είναι πιλωτικό πρόγραμμα, μπορεί να είναι σχέδιο δράσης. Έχουμε 11 αυτή τη στιγμή, νομίζω, σχέδια δράσης μπορεί να είναι και διαδικασία επί παραβάση. Ή διακοπή καταβολής κονδυλίου ή MFF. Ή και αναστολής. Έχουμε, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε εφαρμόσει αυτούς τους μηχανισμούς. Εμείς προσπαθούμε να προσέξουμε, να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα ελέγχου θα λειτουργεί. Έχουμε και τον οργανισμό ελέγχου, ε, τον ΕΦΚΑ, που συνεργάζεται πολύ στενά με τις αρχές των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα αισθήματα ελέγχου ε, χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να τα κάλυψα τα, τα περισσότερα σημεία σας, αλλά ήθελα να επαναλάβω ότι είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε καλύτερα τι έχουμε επιτάπητος, τι, ποιες είναι οι προτάσεις, τι, δια... τι δυνατότητες έχουμε. Είμαστε διαθεσή σας. Γιατί δεν προτείνεται, λέει ο Πρόεδρος, οι ελεγκτικές εκθέσεις να είναι δημόσια διαθέσιμες, των κρατών μελών εννοώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν σας κατάλαβα καλά, Πρόεδρε, δεν δημοσιεύουμε τις εκθέσεις τις ελεγκτικές. Είναι αλήθεια, δεν έχουμε αυτήν την τακτική. Μπορούμε και κλεισμένων των θυρών να το συζητούμε αυτό μαζί σας αλλά κανονικά δεν δημοσιεύουμε τις πληροφορίες σε συγκεκριμένα τμήματα των εκθέσεων αυτών. Γιατί δεν προτείνεται στα πλαίσια της πρότασης αυτού του κανονισμού να είναι δημόσια διαθέσιμες αυτές τις πληροφορίες, λέει ο Πρόεδρος. Ε, πρόεδρε, δεν είναι μέρος πρότασής μας, αλλά ναι, αυτό λέω, λέει ο πρόεδρο. Δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Γιατί δεν κρίθηκε απαραίτητο. Αλλά είναι στα χέρια των συνομοθετών, ε, πρόεδρε. Εντάξει, ικανοποιηθήκαμε. Ευχαριστούμε την Κομισιόν. Yes, indeed. And we will, um, we, we will ask the Commission to uh, make these... Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ε, μελέτες οι οποίες έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τις ε, χρήση συστημάτων, ε, κλειστών συστημάτων τηλεόρασης για την παρακολούθηση των εκφορτώσεων, θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας διαβιβάσει ε, τις σχετικές μελέτες αυτές. Λοιπόν, περνάμε τώρα στα επόμενα σημεία σε ό,τι αφορά τις ε, ε, συμφωνίες αλευτική σύμπραξη της FPA. Λοιπόν, Όπω θα γνωρίζετε, πρόκειται για συμφωνίε τι οποίε έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου τη Ένωση με ε, τρίτε χώρε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με χώρε τη Δυτική Αφρική, αυτέ δηλαδή που θα συζητήσουμε σήμερα. Και οι εν λόγω συμφωνίε επιτρέπουν την αγορά ε, πλεονάζων των ε, αποθεμάτων, αλληλευτικών αποθεμάτων από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και θεωρούνται ω συμφωνίε βιώσιμη αλληλεία. και πραγματικά ελπίζουμε ότι πράγματι είναι συμφωνίε βιώσιμη αλληλεία. Είμαστε λοιπόν αρμόδια από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσουμε αυτέ τι συμφωνίε και συνέχεια να τι εγκρίνουμε. Θα ζητήσουμε λοιπόν τώρα από την Επιτροπή να κάνει μία σειρά από παρουσιάσει των λόγων συμφωνιών. Καταρχήν λοιπόν ζητάμε από την Επιτροπή να μα κάνει την παρουσίαση σε ό,τι αφορά την αλληλεία αλληλευτική σύμπραξη να μα ε, παρουσιάσει τη συμφωνία με το Πράσινο Ακροτήριο. Ο κύριο Μητολίδη, λοιπόν, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει το λόγο. Ε, σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω την τιμή, λοιπόν, να σα ε, εκπροσωπήσω την ε, μονάδα B3 και την κυρία Εντήλη, η οποία δυστυχώ βρίσκεται σε μια αποστολή σε μια πολύ σημαντική χώρα, στο πλαίσιο μια διαπραγμάτευση που γίνεται με εκείνη τη χώρα και γι' αυτό δεν παρευρίσκεται εδώ. Ξεκινάω λοιπόν με τη συμφωνία με το Πράσινο Ακροτήριο του Καμποβέρντη. Ε, και ε, να κάνω ένα σχόλιο εισαγωγικά. Ναι, Πρόεδρε, θεωρούμε πω πρόκειται για συμφωνίε πραγματικά βιώσιμη αλληλεία και έχουμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι είναι βιώσιμε και να διασφαλίσουμε ότι ευθυγραμμίζονται πλήρω με την κοινή αλληλευτική πολιτική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συμφωνία με το πράσινο ακροτήρι. Από τις 20 Μαΐου λοιπόν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, ε, θα αρχίσει να εφαρμόζεται 20 ε, Μαΐου του 2019 ε, στις 20 Μαΐου υπογράφηκε αυτού του ε, έτους λοιπόν και θα τεθεί σε ισχύ από την ε, στιγμή που τα δύο συμβαλόμενα μέρη θα ενημερώσουν το ένα το άλλο σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της εν λόγω συμφωνίας. Ε, πρόκειται για μία ε, συμφωνία αρκετών ετών, μεγάλου δηλαδή διαστήματος, εφιστάμενη συνεργασία με το πράσινο ακροτήριο, η οποία ξεκίνησε αρχικά το 2009 και τώρα καλύπτουμε στρατηγικά, σημαντικές, ε, στρατηγικά σημαντικούς ε, τομείς στο πλαίσιο του ενεργού πρωτοκόλου. Δηλαδή, ε, συμβάλλουμε στην διατήρηση του δικτύου της αλίας των θηνοειδών στον Ατλαντικό. Παρότι μιλάμε μόνο για 750.000 ευρώ ω ετήσια συνεισφορά από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε πω ε, ε, υπάρχει αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη αλληλεία, σε ό,τι αφορά ακριβώ ε, το επίπεδο των αλληλευμάτων. Και θεωρούμε πω το πρωτόκολλο έχει συνάφεια γιατί ακριβώ τοποθετεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στρατηγικά στην ε, εν λόγω περιοχή. Ε, δηλαδή η πρόσβαση στη Δυτική Αφρική είναι πολύ σημαντική για το στόλο μα, ο οποίο αλλιεύει τον θηνοειδή γενικά. Ε, προτείνουμε λοιπόν αλλιευτικέ δυνατότητε για τα σκάφη, τα αλλιευτικά σκάφη, ε, στα ύδατα του Πρασίνου Ακριτηρίου με βάση τι καλύτερε δυνατέ επιστημονικέ πληροφορίες και στο πλαίσιο βέβαια, βέβαια της, ε, της ε, τοπικής, της περιφερειακής ε, ένωσης αλληλείας, της RFMO δηλαδή, συγκεκριμένα του ICAT. Μιλάμε λοιπόν για 8.000 τόνους τόνου και θηνοειδών στα ύδατα του Πρασινού Ακτηρίου και δίνοντας τη δυνατότητα σε αλευτικά σκάφη από την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία να αλλιεύουν εκεί. Και εδώ, όπως είπαμε, εντάσσεται αυτή η συμφωνία στο ευρύτερο δίκτυο αλλίευσης των θηνοειδών στην Δυτική Αφρική. Το λόγο πρωτόκολλο, στο πλαίσιο της χρηματικής αποζημίωσης ε, που προβλέπεται, συμπεριλαμβάνει και υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα δομικά στοιχεία Τη ε, διακυβέρνηση στον αλληλευτικό τομέα στο πράσινο ακροτήρι και ε, θα παίξει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του αλληλευτικού τομέα σε αυτή την ε, χώρα. Η κλαδική λοιπόν στήριξη εδώ προβλέπει ειδικότερα την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, τη βελτίωση της παρακολούθησης και της επαγρύπνησης, βελτίωση της επιστημονικής των επιστημονικών δεδομένων και καλύτερη περιβαλλοντική προστασία ε, και μείωση των σχετικών ταπανών και φυσικά ω συνήθως θα υπάρξει μια κοινή επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί την επιβολή, την εφαρμογή μάλλον του ε, πρωτοκόλου και θα ορίσει τα απαραίτητα βήματα για την επιβολή της νομοθεσίας και όπως είπαμε ακριβώς για την εφαρμογή των εν λόγω ε, ε, τμήματων αυτής της κλαδικής υποστήριξης. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, Κάποιος θέλει το λόγο η, εφόσον αναγκαθεί η έκθεση των συντονιστών, το ΕΛΚΑ θα αναλάβει εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνεχίζουμε τώρα και περνάμε στην Ουινέα Μπισάου. Έχει σχέση, βέβαια. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική μας συμφωνία. Εσείς πάλι έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Προεδρόντο είναι σημαντικό. Η Winner Bissau και το νέο πρωτόκολλο ισχύει προκαταρτικά, προσωρινά, από τον Ιούνιο του 2019. Ήταν ε, μισή χρόνο που μας κράτησε η διαδικασία με διακοπή των αλληλευτικών δραστηριοτήτων εκεί, επειδή ακριβώ είχαν σταματήσει οι διαπραγματεύσει εξαιτία τη πολιτική κατάσταση στη χώρα. Τώρα, θεωρούμε ότι το πρωτόκολλο αυτό είναι ζωτική σημασία για τον ε, ευρωπαϊκό στόλο. Και μάλιστα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν δούμε τη συνολική κατάσταση και την ε, δομή στην ε, Δυτική Αφρική όσον αφορά τον στόλο και του πρασινοκροτηρίου. Εμείς πιστεύουμε ότι με το πρωτόκολλο αυτό έχουμε μια κατάσταση από την οποία έχουν κερδίσουν και οι δύο πλευρές. Ε, θα ισχύει για πέντε χρόνια. Συμπεριλαμβάνεται και νέα κατηγορία μικρών πελαγικών ειδών και η μετάβαση από το σημερινό σύστημα που βασίζεται στην ικανότητα των σκαφών σε ένα σύστημα που έχει να κάνει με το τάξ, που είναι δηλαδή τα νότατα λιεύματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μεγάλη σημασία στην εταιρική σχέση με την Γουινέα Μπισάου και αυτό φαίνεται και από την αύξηση της χρηματοδότησης που είναι 15,6 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 4 εκατομμύρια θα είναι για την στήριξη της ελευτικής πολιτικής στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ελέγξει την εφαρμογή του πρωτοκόλου και να συνεργαστεί στενά με τις αρχές προκειμένου να υπάρξει μία διακυβέρνηση και ένα σύστημα αλληλευτικής διαχείρισης με απόλυτη διαφάνεια υπάρχει το πρόγραμμα στήριξης το οποίο θα καλύψει τις βελτιώσεις στον ελευτικό κλάδο στη χώρα, κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία, την παρακολούθηση, επίσης βελτίωση της επιστημονικής ικανότητας και κάτι άλλο σημαντικό που πιστεύουμε εμείς ότι παίζει σημαντικό ρόλο είναι η δική μας συνεισφορά στην διατροφική ασφάλεια στη χώρα. Και αυτό επιτυχάνεται επειδή προβλέπουμε υποχρεωτικές εκφορτώσεις στη χώρα για τον τοπικό πληθυσμό. Θα υπάρξει μεικτή επιτροπή, η οποία θα παρακολουθήσει από κοντά και θα ελέγχει την εφαρμογή της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μητολίδη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις προσπάθειες που έκανε προκειμένου η συμφωνία αυτή να καταλήξει θετικά. Τόσο η συμφωνία αυτή όσο και η προηγούμενη που εξετάσαμε με το πράσινο ακροτήρι είναι συμφωνίες πολύ σημαντικές για τα καταψυχτικά των οθυρικά και για την Ισπανία, από τη χώρα των Βάσκων, που, που έρχομαι εγώ για παράδειγμα, πρέπει να ξέρετε ότι δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης εκεί όπου πηγαίνουν και αλλιεύουν. Άρα απασχόληση, πλούτο και βέβαια και στην Ευρώπη. Στηρίζουμε, εννοείται, και πράγματι είναι μια σημαντική συνεισφορά για τη διατροφική ασφάλεια στην περιοχή, μια που υπάρχει υποχρέωση για ποσόστοση εκφορτώσεων η οποία θα προορίζεται για τον ντόπιο πληθυσμό. Ευχαριστώ, κύριος Γκριζάλης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εννοείται, και εγώ θέλω να στηρίξω την συμφωνία αυτή, είμαι από τη Γαλλικία και η αλία είναι κάτι παραπάνω από ένα τρόπο ζωής για μας. Στηρίζουμε πάνω απ' όλα για τη συμφωνία με τη Γουενέα Μπισάο είναι κάτι που περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Ισπανία και στη δικιά μου την περιφέρεια αλλά και σε ολόκληρη την Ισπανία. 16 σκάφη από την Γαλλική εκδοδόση, από την Ισπανία ολόκληρη θα αποφεληθούν. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό νέο όχι μόνο για τον αλληλευτικό στόλο της Γαλλικίας και της Ισπανίας, αλλά και γενικότερα για τη διεθνή συνεργασία με μια υποανάπτυξη χώρα όπως είναι Γουινέα Μπισάου. Στηρίζω λοιπόν και προσθέτω ότι τα νέα μοντέλα που αναφέρονται στο πρωτόκολλο, για παράδειγμα για την εξασφάλιση της διατροφής ε, την χώρα ή για το ότι θα μπορούν να είναι περισσότεροι ναυτικοί πάνω στα σκάφη αυτά από τον τόπιο πληθυσμό είναι θετικά. Χαίρομαι λοιπόν για την συμφωνία αυτή και θα ε, συνεχίσουμε να την ελέγχουμε. Είναι πάντως σημαντική και θα τη στηρίξουμε. Ευχαριστούμε. Περίρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για αυτή την παρουσία σε ό,τι αφορά αυτή τη διαπραγμάτευση η οποία έγινε, θεωρούμε πως ε, έγινε με έναν συντονισμένο λόγο και θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι ήταν δυνατόν να υπάρξει μια ευθυγράμμιση, μια προσέγγιση μεταξύ των ε, δύο συμβαλωμένων μερών, ειδικότερα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ελήφθησαν δηλαδή περισσότερο υπόψη οι ανησυχίες των αρχών ε, της Γουινέα Μπισάου. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τη Γουινέα Μπισάου το 2016, ε, δηλαδή πριν από τρία χρόνια και παραπάνω, για να παρακολουθήσουμε ακριβώς την εφαρμογή της προηγούμενης συμφωνίας, για να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι ελλείψεις ακριβώς σε ό,τι αφορά την ε, παροχή αυτής της κλαδικής υποστήριξης που έχουμε στη Γουινέα Μπισάου. Είναι λοιπόν θετικό το γεγονό ότι ορισμένε από αυτέ τι ανησυχίε ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την τεχνική υποστήριξη, την συνεργασία στο επίπεδο ε, των ελέγχων, τη επιθεώρηση ε, και ούτω καθεξή ελήφθησαν υπόψη με αποτέλεσμα να βελτιωθούν ακριβώ οι δυνατότητε που έχει αυτή η χώρα σε αυτού του τομεί. Και επίση είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει πιο σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι πέραν από την παροχή χρηματικών πόρων για την κλαδική υποστήριξη, να δώσει περισσότερους, ε, περισσότερες δυνατότητες για την απορρόφηση των συγκεκριμένων πόρων. Δηλαδή να δώσει περισσότερες ε, δυνατότητες, περισσότερα εργαλεία στις αρχές της Γουινέα Πισάου, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την απορρόφηση των λόγω, ε, την λόγω χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά την κλαδική υποστήριξη. Για παράδειγμα, στο επίπεδο των υποδομών. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι μία από τις ανησυχίες των αρχών της Γουινέα Πισάου και μια πραγματικά δίκαια ανησυχία είναι ότι ε- ε- ε- επιβάλλεται αυτή η υποχρέωση εκφόρτωση στου λιμένε τη εν λόγω χώρε. Η Επιτροπή λοιπόν λέει ότι ναι, θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση εκφόρτωση, αλλά δεν υπάρχουν οι απαραίτητε υποδομέ στου λιμένε τη χώρα για να εφαρμοστεί αυτή η υποχρέωση. Άρα λοιπόν. Εδώ βλέπουμε μια αδυναμία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα σε τρει τρεις δεκαετίες οι οποίες συνάπτονται με την Γουενέα Μπισάου να εξασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις οι οποίες πραγματικά θα επιτρέπουν σε αυτή τη χώρα να προβαίνει στην επιβολή των υποχρεώσεων εκφόρτωσης. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή αυτό που δεν κατάφερε να κάνει μέσα σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια να φροντίσει να μην συνεχίζει να αποτυγχάνει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια και νομίζω πως θα πρέπει να αποτελέσει και στο μέλλον ε, ζήτημα που θα απασχολήσει και εμά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρέπει να αναφερθεί και μέσα σε αυτή την έκθεση που θα προετοιμάσουμε ακριβώ σε σχέση με την Ελόγω Συμφωνία. Να κάνουμε δηλαδή κάποιε συστάσει σε αυτή την έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να βελτιώσει προ αυτή την κατεύθυνση και στα διάφορα επίπεδα τη συμφωνία με την Γουινέα Μπισάου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, εγώ ήθελα να επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντική η συμφωνία μετά την Μαυριτανία και το Μαρόκο είναι ο τρίτος πιο σημαντικός εταίρος. Είχαμε αναστείλει τη συμφωνία 24 μηνών, εγώ ρωτούσα συνέχεια. Έκανα συνέχεια ερωτήσεις προς την Κομισιόν και νομίζω από τις 15 Ιουλίου αλλιεύουμε. Για εμάς μιλούμε για πάνω άνω των 50 σκαφών και 16 από την Γκαλήθια. Ε, επίσης υπάρχει και ο στόλος των κεφαλόποδων, ε, ο οποίος έχει ζωηρό ενδιαφέρον. Επίσης να σας πω, Πρόεδρε, ότι ο κύριος Βαντάλεν θα είναι ο εισηγητής του ΕΛΚ και μου ζητά να υπογραμμίσω τη σημασία της συμφωνίας αυτής για τον ευρωπαϊκό στόλο αλλά και για τον στόλο και την ίδια τη χώρα της γωνιάς Μπισάου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μιχαηλίδη, ε, σχετικά με τις παρατηρήσεις των μελών, κύριε Μητολίδη, στο συγγνώμη, ε, επανεξετάσαμε την ΚΑΠ ε, του 2014 ε, για να την καταστήσουμε βιώσιμη. Εσείς είχατε υπογραμμίσει διάφορες ε, διευθετήσεις ε, των συμφωνιών που συμμετείχαν στο πλαίσιο αυτό. Εσείς παρατηρείτε, σημειώνετε κάποια διαφοροποίηση για το πώς διαπραγματευόμαστε αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας σήμερα σε σχέση με το πώς το κάναμε πριν από 10 χρόνια. Επίσης, είμαστε σε ανταγωνισμό με την Κίνα και πολλούς άλλους στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών. Πώς τις κερδίζουμε, επειδή δίνουμε περισσότερα χρήματα ή επειδή προσπαθούμε να καλύψουμε κοινώ επωφελή ζητήματα και για εμάς και για τη χώρα με την οποία διαπραγματευόμαστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σημειώσαμε τα εξαιρετικά σημαντικά σχόλια και παρατηρήσεις των μελών που μας υποβάλλουν ε, σχετικά με τη συμφωνία. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της συμφωνία αυτής για τον Ευρωπαϊκό Στόλο, το είπατε. Σημειώνουμε επίσης τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος για τη Γουινέα Μπισάου, για την έλλειψη εξοπλισμού, για τα όσα έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το νέο πλαίσιο των συμφωνιών για τη βιώσιμη αλληλεία και ο νέος περίφημος ΣΜΕΦ κανονισμός μας έχουν βοηθήσει να κινηθούμε σημαντικά προς τα εμπρός για τον τρόπο με τον οποίο λεμανόμαστε και εμείς και οι εταίροι μας την υλοποίηση. Νομίζω ότι το είχαμε αναφέρει και στην Κοινή Επιτροπή και θα κοιτούμε με έντονο ενδιαφέρον στα θέματα της υλοποίησης εποφελούς και για τα δύο μέρη και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε γενικό επίπεδο για το τι κάνουμε στα πλαίσια αυτών των ε, εταιρικών συμφωνιών βιώσιμης αλίας, έχουμε απομακρυνθεί από σφάλματα του παρελθόντος και γι' αυτό μετά από μακρά διαδικασία προπαρασκευαστική και συζητήσεων διαπραγματεύσεων μεταξύ δύο, ε, των δύο συνομοθετών έφτασε αυτός ο κανονισμός ΣΜΕΦ και οι κατευθυντήριες αρχές μας, η βίβλος μας είναι η κοινή αλληλευτική πολιτική η οποία με σαφήνεια λέγει ότι καλούμαστε μεταξύ άλλων να επιτύχουμε περιβαλλοντική ιδιωσιμότητα οικοδομούμε τις παρεμβάσεις μας στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου δεν πάμε εκεί να αφαιρέσουμε πόρους που δεν υπαρκούν. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονάσματα επί τη βάση και του ούγκλος και των διεθνών συμφωνιών είμαστε απολύτως διαφανείς για το σύστημά μας. Όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορίε, στις πληροφορίες, τα δεδομένα των οποίων βασίζουμε τις αποφάσεις μας και για το πώς αφαιρούμε τα αποθάματα αυτά από τα ύδατα των παρακτήων κρατών και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι κάνουν άλλες χώρες διεθνώς, οι οποίες δεν ακολουθούν αναγκαστικά την ίδια προσέγγιση. Ακολουθούμε επίσης μια προσέγγιση απολύτως κατά των διακρίσεων για την πρόσβαση των δικών μας στόλων, του δικού μας κλάδου στις αγορές. Έχουμε πολύ στοχευμένες ιδέες και πολύ καλά επιλεγμένες για το τι θέλουμε, πώς θέλουμε να βοηθήσουμε τις παράκτιες χώρες, ιδιαίτερα στα θέματα παρακολούθησης και ελέγχου, επιστημονικών συμβουλών, στα πλαίσια της προσπάθειάς μας επίσης της καταπολέμησης της παράνομης αλίας. Επομένως πραγματικά θεωρούμε ότι είμαστε οι good guys εδώ, είμαστε οι καλοί στο πλαίσιο αυτό. Εξαιρετική η σύνοψή σας, λέει ο Πρόεδρος, εξαιρετική. Ε, να πάμε στο τρίτο σημείο υπό τη δέσμη αυτή και εδώ μιλούμε για την Κάμπια, σας ξαναδίνω το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, το τελευταίο λοιπόν που θέλαμε να σας παρουσιάσουμε είναι η συμφωνία με την Κάμπια. Η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γκάμπια είναι από τα πιο παλαιά τέκνα το 87 είχε ξεκινήσει η προσπάθεια αυτά και το τελευταίο πρωτόκολλο το 96. Τον Οκτώβριο του 18 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με η νέα συμφωνία και νέου πρωτοκόλλου με τη χώρα απολύτως ευθυγραμμισμένου με τους ε, αρχές και τους στόχους της ΚΙΑΠ. Η νέα συμφωνία ενέχει νέες δυνατότητες για τα θηνοειδή, τον ε, γάδο ε, και τα παραγατιάρικα χρησιμοποιήσαμε, αν θέλετε, την πυθό μας, ώστε η χώρα η συγκεκριμένη να γίνει μέλος της ICAT, καθότι αυτό είναι νομική προϋπόθεση του ΣΜΕΦ, ο οποίος προβλέπει ότι οι εταίροι πρέπει να είναι μέλη των περιφερειακών οργανώσεων αλίας. Και η νέα συμφωνία επίσης προσπαθεί να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει παράνομη λαθρέα και άναρχη αλία, να χρησιμοποιήσει μόνο το πλεόνασμα των πόρων και να βασίζεται μόνο στις βέλτιστες επιστημονικές συμβουλές για την καλύτερη αλληλευτική διαχείριση. Η νέα συμφωνία επίσης θα είναι μέσον υποστήριξης βοήθειας της τοπική οικονομίας, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης θεωρούμε και θα βοηθήσει και στη σταθεροποίηση της νέας πολιτικής ηγεσία στη χώρα. Ε, Ευχαριστούμε, κυρία Ρούτς. Ακόμα και αν η συμφωνία προβλέπει δυνατότητες αλλιές, προβλέπει επίσης ε, και για τα σε μεγάλο βάθος πελαγιακά είδη και αυτό θέτει ερωτήματα. Λίγο πολύ πήρα απάντηση για την τοπική αλία, αλλά θέλω να ρωτήσω και το εξή. Πώ η τύποση μπορεί να διασφαλίσει ότι τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ταράζουν την τοπική αλία και οι τοπικοί πληθυσμοί έχουν ε, ερωτηθεί στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Τώρα όσον αφορά τις διατάξεις, οι διατάξεις της πρότασης αρκούν για την συλλογή των ε, δεδομένων για την αλία στο θαλάσσιο χώρο και κυρίως για τα είδη. Η επιστημονική αξιολόγηση από την άλλη έχει δώσει αρκετά αποτελέσματα που να δείχνει ότι ε, τι γίνεται με τα ίδια αυτά σε μεγάλο βάθος τα πελαγιακά και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Άλλος κανείς. Παρακαλώ. Για την απάντηση τότε. Μερικές φορές έχει ακουστεί ότι φτάνει ο ευρωπαϊκός στόλος και ότι αυτοί που είναι στην εξουσία σε τοπικό επίπεδο δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Εσείς μας υπόσχεστε ότι αυτό δεν συμβαίνει πια, ότι τους λαμβάνουμε υπόψη, τον κόσμο δηλαδή γενικά. Θα απαντήσω όσον αφορά τα πελαγιακά είδη. Πρέπει να ξεκινήσουμε την εξάντε αξιολόγηση για τον μπακαλιάρο της Ενεγάλης. Να υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν αυτά τα είδη. Ο τοπικός πληθυσμός, δεν υπάρχουν βέβαια τοπικά αλής ε, για αυτά τα είδη. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό είναι ένας λόγος που εμείς πηγαίνουμε εκεί με τον Οθυρικά, για παράδειγμα. Αλλιώς δεν θα το είχαμε κάνει αν υπήρχαν εκεί ε, τοπική αλύση. Πώς λοιπόν θα διασφαλίσουμε, λέτε, την βιώσιμη αλία. Πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι μπορούμε, γιατί υπάρχουν επιστημονικές εκθέσεις από τη ΣΕΚΑΦΑ, που είναι ο οργανισμός που δίνει επιστημονικές συμβουλές, που λέει ότι είναι βιώσιμη η αλία του γάτου και από την άλλη μεριά Υπάρχει και η Επιστημονική Επιτροπή και η Μικτή Επιτροπή Ελέγχου. Εδώ δεν θα έχουμε μόνο αυτήν την ε, Μικτή Επιτροπή Ελέγχου, αλλά θα έχουμε και την Επιστημονική Επιτροπή, προκειμένου να ελέγχεται η υλοποίηση των συμφωνιών ε, αυτών, που είναι μικτές, όπως και στην περίπτωση της Γκάμπια. Οι ελίς πρέπει να έχουν έναν επιστημονικό παρατηρητή στα σκάφη τα οποία αλλιεύουν γάδο στη χώρα. Επιπλέον έχουν και την υποχρέωση για ένα ποσοστό τοπικών ε, ναυτών να έχουν στα σκάφη τους. Ευχαριστούμε. Άλλος. Ωραία. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω το ότι είμαστε καλοί ε, να είναι κάτι ουδέτερο το οποίο να μας αφορά όλους. Ουδέτερο κατά το φύλλο. Καλή και καλές. Μια μικρή διακοπή να δούμε αν για το επόμενο θέμα είναι εδώ εκπρόσωποι της Επιτροπής. Okay, Τρία λεπτά διακοπή. Στις και πέντε θα αρχίσουμε και πάλι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 Με στέλνουν σε διάφορα χωρίς να υπάρχει λόγο. Ε, δεν είναι κανείς το Δεν είναι το Και μου το Και μετά μου λένε αφού δεν σήκει δεν κάνεις αυτό γιατί το μόνο που Ελλήνης είναι διαβρετανά. Καινούργια.

εγώ ψάχνω κάποιον για τα διεθνή θέματα, για το UN και τέτοια να βοηθήσει.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 Uh, λοιπόν, χτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε εκτάκτος μέτρα για την ε, διατήρηση του γάδου στην Ανατολική Βαλτική θάλασσα. Υπήρχε έκθεση του Μαΐου του ICS που έλεγε ότι τα αποθέματα γάδου μειώνονται σημαντικά. Οπότε, κύριε Φρύς, έχετε το λόγο για να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Uh, για αυτή την παρουσίαση που θα κάνω σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην ε, Βόρειο Θάλασσα, στον Ατλαντικό, στη Βαλτική και όπως ε, ακούσατε ή μάλλον είπατε ο ίδιος, ε, υιοθετήσαμε κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά με την Ανατολική Βαλτική για ορισμένα μέτρα ...και την καταπολέμηση τη παράνομη λαθρέα και άναρχη ε, αλληλεία με βάση επιστημονικά δεδομένα που λάβαμε στα ε, τέλη Μαΐου. από το Συμβούλιο ISIS, την περιφερειακή δηλαδή οργάνωση που αναφέρει και κοινοποίησε σε εμά και στις ενδιαφερόμενες ε, χώρες ότι τα αποθέματα του τόνου στην ε, Ανατολική Βαλτική μειώνονταν εδώ και χρόνια, αλλά δηλαδή πραγματικά έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο επίπεδο. Εξαιρετικά δηλαδή κακή κατάσταση. Και ε, θεωρείται πως η βιομάζα πλέον των αποθεμάτων το spawning biomass, ε, δηλαδή τα, ο αριθμός των ηχθείων που είναι απαραίτητος ώστε να μπορεί να πολλαπλασιάζεται το απόθεμα, είναι πλέον, δεν, δεν πληρείται πλέον, δεν είναι επαρκής. Κατά συνέπεια λοιπόν η ικανότητα του αποθέματος ε, τόνου βρίσκεται πλέον σε, κίνδυνο. Ο, οι λόγοι δεν είναι σαφείς, αλλά είναι πιθανό ότι οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, δηλαδή πολύ απλά μόλυνση της Βαλτικής και σε αλλαγές οικοσυστήματος ε, οι οποίες οφείλονται ε, πιθανότατα στην κλιματική αλλαγή. Και βέβαια η αλληλευτική δραστηριότητα επιβάλλει πιέσεις ε, στα, στα, αποθέματα. Δηλαδή δεν είναι υπεύθυνη η αλληλεία για τη μείωση του αποθέματος, αλλά συμβάλλει στη μείωσή του. Άρα λοιπόν ε, βρίσκεται πλέον σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα η, βιώσιμη, ε, η βιομάζα του, του αποθέματος από τότε που έχει αρχίσει να καταγράφεται. Ε, έχουμε λοιπόν τώρα την έναρξη της, της έκτακτης διαδικασίας όπως ε, προβλέπεται ε, στον κανονισμό για την κοινή πολιτική και ουσιαστικά αυτά τα έκτακτα μέτρα επιβάλλουν άμεση απαγόρευση της αλληλείας του συγκεκριμένου αποθέματος και με αυτόν τον τρόπο η επιβολή των μέτρων γίνεται με τον όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο δηλαδή επιτρέπεται η αλληλεία άλλων κατηγοριών που είναι σχετικές, δηλαδή ε, παράκτη αλληλεία, ριχά δηλαδή ύδατα, ε, στα, στα μέσα της ε, Βαλτικής, στην περιοχή 24 συγκεκριμένα, μετά παρεμπίπτωτα ε, αλλιεύματα τόνου, δηλαδή από άλλα πελαγικά είδη που αλλιεύουν άλλους, άλλα σκάφη με άλλο στόχο. Και επίση αλλιευτική δραστηριότητα μικρού μεγέθου ε, σκαφών μέχρι ενό σημείου. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν ε, πολύ χαμηλέ ποσοστό σε ό,τι αφορά την αλληλεία γάδου σε, αυτόν τον, σε αυτή την περιοχή και αυτές είναι εξαιρέσεις που έχουμε προβλέψει. Ναι, το ΆΣΙΣ ε, έχει ε, κάνει κάποιες συστάσεις ε, από το 2020 και μετά και προτείνει λοιπόν να είναι πολύ περιορισμένη η αλία γιατί πραγματικά οι προοπτικές του συγκεκριμένου αποθέματος δεν είναι καλές του γάδου. Οπότε τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι η καλύτερη οδός σε προληπτικό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να επιτρέψουμε την αποκατάσταση του συγκεκριμένου αποθέματος. Πρόεδρος. Ε, θα ακούσουμε και ποιοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο, αλλά να ρωτήσω και εγώ. Ποιο είναι ο αριθμό ε, των αλλιέων που θίγονται άμεσα από αυτή την επιβολή τη απαγόρευση. Και σημαίνει ότι θα πρέπει να πάυσουν την αλληλευτική του δραστηριότητα ή θα έχουν τη δυνατότητα να ε, ξεκινήσουν την αλληλεία σε άλλη περιοχή. Ε, να δώσω το λόγο καταρχήν στον κύριο Γκίργε συνέχεια στους υπόλοιπους ομιλητές η αλληλεία ε, στην Βαλτική ε, προφανώς έχει μια συγκεκριμένη σοβαρότητα γιατί ε, καταρχήν δεν έχουμε την ίδια αξιοποίηση αυτών των αλληλευτικών αποθεμάτων από τις χώρες της ε, Βαλτικής. Ε, κυρίως δηλαδή εδώ θίγεται η Λιθουανία από την επιβολή αυτών των μέτρων και με βάση τα στοιχεία μας γύρω στο 1 τέταρτο του αλληλευτικού στόλου της Λιθουανίας εξαρτάται από την αλλήλευση του γάδου. Και σε ορισμένε περιοχέ μιλάμε για το 90% του αλευτικού στόλου το οποίο επιτίθεται σε αυτή τη δραστηριότητα. Οπότε εδώ θα υπάρξει σημαντικό αντίκτυπο. Ε, ε, αντίστοιχο, αντίκτυπο θα έχουν αυτά τα μέτρα για τον ε, πολωνικό ε, στόλο. Μπορώ να σα δώσω ε, και πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά το τμήμα του αλευτικού στόλου που θίγεται από τι διάφορε χώρε. Αν θέλετε, μπορώ να το εμβάσω στην γραμματεία. Δεύτερη ερώτηση του Προέδρου. Οι εν λόγω λοιπόν στόλοι απλώς δεν θα μπορέσουν να αλλιεύουν από εδώ και στο εξή ή θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν αλλού την ελεύθερη τους δραστηριότητα. Απάντηση. Ε, δεν είναι προφανέ ότι όλοι αυτοί οι στολοί, όλα αυτά τα σκάφη θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν αλλού. Δηλαδή, ένα σημαντικό αριθμό, ναι, δεν θα μπορέσει να, να λάβει δράση. Να, να, να ξεκινήσει δηλαδή αλληλεία. Και ε, το πιο σημαντικό είναι ότι μακροπρόθεσμα ε, υπάρχει ε, ζήτημα γιατί υπάρχει ε, τμήμα του ελευτικού στόλου που ειδικεύεται στην αλληλεία αυτού του είδους και βλέπουμε ότι το εν λόγω απόθεμα για αρκετά μεγάλο διάστημα δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποκατασταθεί. Με βάση τα όσα προβλέπει τώρα ο σχετικός κανονισμός, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν χρηματοδοτική υποστήριξη στους αλληλείς εκείνους που θίγονται ακριβώ από τέτοιου είδου ε, προσωρινά μέτρα απαγόρευση τη αλληλεία. Ε, υπάρχουν αυτέ οι δυνατότητε για τα κράτη-μέλη, οι οποίε δεν έχουν αξιοποιηθεί ε, πλήρω. Οπότε, στο πλαίσιο του κανονισμού για το EMFF, το Ταμείο δηλαδή Θάλασσα και Αλληλεία, υπάρχει δυνατότητα και έχουμε έρθει σε επαφή με αυτέ τι χώρε έτσι ώστε να αξιοποιήσουν αυτέ τι δυνατότητε εφόσον το επιθυμούν. Γιατί την απόφαση για την χορήγηση τέτοιου είδου υποστήριξη δεν την λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ στι Βρυξέλλε, αλλά τη λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Εδώ. Ε, να ξέρετε ότι η δανέζικη συνδιαλέγει. δεν ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Ονομάζομαι Σάνμπερκ, είμαι από τη Δανία, ναι. Και σίγουρα είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, γιατί εγώ είμαι από την χώρα αυτή στην οποία υπάρχουν επιπτώσεις από αυτή την απόφαση. Είναι μια απόφαση που θα επηρεάσει εκατοντάδες οικογένειες και τον τρόπο ζωής τους. Πρέπει να πω ότι αν κοιτάξουμε την έκθεση της ISIS, έχουν εκτιμήσει ότι αν υπολογίσουμε ολόκληρα τα αποθέματα, μόνο 4% ε, θα είναι επιπτώσεις το 2020. Οπότε σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στην Ανατολική Βαλτική, αλλά αυτό που θα έπρεπε να δείτε είναι ότι κάποια κομμάτια αυτής της περιοχής, αν δείτε το δυτικό μέρος του τμήματος 24, εδώ το ποσοστό θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι ναι, φυσικά και πρέπει να προσέξουμε ε, το γάδο στο ανατολικό τμήμα, αλλά είναι πολύ μεγάλη η περιφέρεια που περιορίζεται και θα έπρεπε να το έχετε υπόψη σας εξετάζοντας τις επιπτώσεις όχι μόνο τώρα, αλλά και μετά το 2019, γιατί θα επηρεαστούν, όπως σας είπα, Πολύ αλής στην περιοχή. Σας ζητώ λοιπόν να κοιτάξετε αυτήν την υποδιέρεση 24. Ε, πρόεδρος, ε, πρόκειται για έκτακτα μέτρα, έτσι, για έξι μήνες. Η πρόταση θα είναι από πλευρά των επιστημόνων ότι δεν θα υπάρξει ποσόστοση για το μέλλον. Δεν πρόκειται για μια μόνιμη, για μόνιμα μέτρα είναι μόνο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου τα αποθέματα να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι. Ναι, ναι, όντως, πρόκειται για έκτακτα μέτρα τα οποία ισχύουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τότε θα αρχίσει να ισχύει η νέα ρύθμιση για τις ελλειφτικές δυνατότητες. Θα τα αποφασίσει το Συμβούλιο, όπως ξέρετε, το Δεκέμβριο. Και οι επιστήμονες μας λένε ότι αν σταματήσουμε την αλίευση τώρα, θα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις, δηλαδή περιμένουμε ότι θα υπάρξει κάποια μικρή έστω βελτίωση που αξίζει τον κόπο. Εμείς προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα μέτρα έτσι ώστε να είναι αναλογικά, να περιορίσουν δηλαδή τις επιπτώσεις σε ε, αλείς οι οποίοι δεν είναι αλείς γάδου με τις τρεις εξαιρέσεις που σας είπα στην αρχή γιατί ίσως τότε να ήταν δυσανάλογα τα μέτρα. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε γενικά ε, τους αλείς, ακόμα και αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο. Τώρα για την υποδιέρεση 24 περίπου 75% των αλλιευμάτων σε αυτή την περιοχή είναι από τα ανατολικά αποθέματα, τα αποθέματα στα οποία αναφέρεται το μέτρο. Οπότε αν πάρετε μια αρχή προφύλαξης και την εφαρμόσετε, αυτό πρέπει να κάνετε. Και για μας αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Τα έκτακτα μέτρα καλύπτουν το 24, 25 και 26 και τις τρεις αυτές υποδιαιρέσεις. Τίποτα πιο βόρεια όπου υπάρχουν ε, λίγα αποθέματα. Θέλαμε στοχευμένα να είναι τα μέτρα μας. Και στην υποδιέρεση 24 προσπαθούμε να αποκλείσουμε με λειτουργικό τρόπο, με ελεγχόμενο τρόπο να αποκλείσουμε αυτούς που βρίσκονται κοντά στις ακτές ή σε πολύ ρηχά ύδατα. Πρέπει να γίνει βέβαια παρετέρω συζήτηση με ειλικρίνεια και να αναλύσουμε τις προτάσεις για το 2020 και μετά, όπως σωστά είπατε. Οι συζητήσεις θα γίνουν στο Συμβούλιο και εκεί θα απαρθούν τελικά οι αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μια μικρή παρατήρηση επιτρέψτε μου ακόμα. Μα στο δυτικό κομμάτι του 24 δεν είναι το ίδιο με το ανατολικό. Εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω δεν είναι ο γάδος στο δυτικό τμήμα. Και έπειτα από αυτά που λέτε, όλα αυτά θα επηρεάσουν πάρα πολύ κόσμο για ένα 4%. Μα αναρωτιέμαι, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Τα επόμενα χρόνια και αλλού στην Ευρώπη θα έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα έπρεπε να το δούμε συνολικά, γιατί ίσως μπορούν να γίνουν και άλλα πράγματα. Όχι απλώς να κλείνουμε μια περιοχή και να απαγορεύουμε στον κόσμο να λιεύει, οπότε δεν μπορεί να ζήσει από αυτή τη δραστηριότητα. Θέλω να υποστηρίξω κατηγορηματικά τα όσα είπε ο ενός συνάδελφου. Δηλαδή δεν θα πρέπει να εξετάσουμε μόνο το ζήτημα του γάδου, αλλά και το τι αυτό θα σημάνει ε, σε ό,τι αφορά τη δυτική περιοχή της ε, Βαλτικής, καθώς όσοι δραστηριοποιούνταν εκεί στην Ανατολική θα μεταφερθούν στη δυτική περιοχή. Αυτό λοιπόν θα έχει επιπτώσει κατευθείαν και στη δυτική πλευρά της ε, Βαλτικής. Και εδώ λοιπόν Έρχομαι σε αυτό που ε, είπε ο συνάδελφο, δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχουμε αντιμετωπίσει διαφοροποιημένα την περιοχή 24. Με αυτόν τον τρόπο θα, μειώσαμε, θα μειώναμε τι δυνατότητε άσκηση περισσότερων αλληλευτικών πιέσεων στον ε, Γάδο και στη δυτική πλευρά τη ε, Βαλτική. Και σε ό,τι αφορά αυτά που είπε πρόσωπο τη Επιτροπή, διαρωτώ με σε ό,τι αφορά την, και την τήρηση τη αναλογικότητα, αλλά ε, και το κατά πόσο, για παράδειγμα, υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση βάρο των σκαφών εκείνων τα οποία έχουν μεγαλύτερο μέγεθο. Ε, ε, πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή το έχει διασφαλίσει αυτό από άποψη, για παράδειγμα, τήρηση πράγματι τη αρχή τη μη διακριτική μεταχείριση. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει, άμα περάσει από το ανατολικό τμήμα στο δυτικό, πιέζεται περισσότερο το δυτικό τμήμα. Τι έχετε να πείτε, είναι κάποιες χώρες που πλήττονται περισσότερο από κάποιες άλλες, σωστά. Ναι, ευχαριστώ για το θέμα αυτό, για την αλλαγή αυτή προς τα αποθέματα δυτικά. Όπως γνωρίζετε, έχει τη δικιά του ιστορία το απόθεμα δυτικά, άλλου είδου προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις κλιματικές συνθήκες μεταξύ άλλων που τα αποθέματα εκεί υποφέρουν διαφορετικά από ό,τι στο ανατολικό τμήμα. χρησιμοποιήθηκε πολύ το απόθεμα του γάδου εκεί. Οι ποσοστώσεις όμως υπάρχουν και δεν είναι δυνατόν ένα αλιές που έρχεται από μια άλλη περιοχή να βρεθεί στο δυτικό τμήμα της Βαλτικής και να ψαρεύει εκεί, πρέπει να έχει ποσόστοση. Οι ποσοστώσεις ρυθμίζονται με συγκεκριμένους κανονισμούς και ευθυγραμμίζονται με τις αρχές της προφύλαξης στα δυτικά αποδέματα. Αν έχετε ε, δηλαδή ποσόστοση μπορείτε να λιεύετε εκεί. Αν δεν έχετε ποσόστοση δεν μπορείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα έρχομαι στην ερώτησή σας για το πώς να διαχειριστούμε το κομμάτι 24. Με συμβουλή του ISIS εμείς πήραμε αυτά τα μέτρα, συμβουλευτήκαμε και τον ISIS πέρα δηλαδή από την έκθεσή τους. Πραγματικά προσπαθήσαμε και διαφορετικά. Αλλά είναι δύσκολο λειτουργικά να διακρίνει κανείς το δυτικό από το ανατολικό τμήμα. Πιστεύουμε ότι αν μπορούμε έστω και λίγο να βελτιώσουμε το μέγεθος των αποθεμάτων, πρέπει αυτή την ευκαιρία να την χρησιμοποιήσουμε. Και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κλείσουμε ολόκληρη την περιοχή. Ευχαρίστως όμως να κοιτάξουμε μαζί γραμμή προς γραμμή την επιστημονική έκθεση. Ζητήσαμε συμβουλές, τις αναλύσαμε, τα συζητήσαμε με ειδικού στην Αλία στις ενδιαφερόμενες χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί κατέληξε και γι' αυτό ενέκρινε αυτό που ενέκρινε χτες. Ένα σύντομο δεύτερο ερώτημα. Οι ποσοστώσει που έχουν για παράδειγμα η Πολωνία και η Λιθουανία σε ό,τι αφορά το γάδο στην ε, δυτική ε, πλευρά τη Βαλτική έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο ή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ακριβώ για να αμβληθούν οι πιέσει από τι ελευθερικέ δραστηριότητε που θα μετατοπιστούν. Κοιτάξτε, να το ελέγξω για να είμαστε απόλυτα σίγουροι, αλλά νομίζω ότι η ποσόστος του δυτικού γάδου, βέβαια είμαστε στα μέσα του έτους, σημειώστε, έχουμε ακόμα μισή περίοδο μπροστά μας, και δεν νομίζω ότι οι αλείς που θα μπορούσαν να επιφαληθούν της ποσόστοσης αυτής θα μπορούσαν να εμπέσουν στην τρέχουσα περίοδο. Πάντως, στη Δυτική Βαλτική συνήθως ήταν χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Σουηδία που εποφελούνται και το ανατολικό τμήμα της Βαλτικής, Πολωνία, Λιθουανία και άλλες χώρες με, μια μικρή συμμετοχή ποσόστοσης εκατέρωθεν στα δύο αυτά μέρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη δυνατότητα, αλλά δεν μπορώ να είμαι 100% βέβαιος αυτή τη στιγμή. Για μετακίνηση δηλαδή εσείς στο άλλο διαμέρισμα. Να το ξαναελέγξω και να σας δώσω ακριβέστερα στοιχεία. Ε, θα σας... Ήμασταν υπόχρεοι, λέει ο πρόεδρος. Ε, παραλιεύματα μέχρι 10% είναι για το γάδο. και πώς το ε, ελέγχεται αυτή την ποσότητα του παραλίευματος. Ναι, κοιτάξτε, εδώ είμαστε σε μία από τις τρεις εξαιρήσεις μικρής κλίμακας αλίας και συγκεκριμένα μεγέθη σκαφών και είναι θέμα αλληλευτικών ελέγχων που εξασφαλίζουν τα κράτη-μέλη. Καθένα από τα οποία έχει τις δικές του ελεγκτικέ αρχές και μηχανισμούς και εξασφαλίζεται έτσι ότι όλα αυτά παρακολουθούνται. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε ποσόστοση, ούτως ή άλλως. Άρα τελευταία διαφημιστική από πλευρά μου λέει ο πρόεδρος έχετε εισαγάγει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Θα επεκταθούν αυτά στο νέο έτος, θα έχουμε απαγόρευση για το γάδο. Αν δεν είχατε εισάγει τα μέτρα αυτά, τι θα είχε γίνει με το απόθεμα. So, in, in the now Κοιτάξτε, σε ένα τέτοιο υποθετικό σενάριο, κατά το οποίο δεν θα είχαμε υιοθετήσει τις ρήτρε αυτές όπως τις έχετε μπροστά σας και αν δεν είχαμε υιοθετήσει τις επιστημονικές ε, συμβουλές θα είχαμε μείωση της βιομάζας του αποθέματος. Μας λένε οι επιστήμονες ότι το απόθεμα αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία για να αναπαραχθεί. Κυρίως μιλούμε για νεαρά άτομα τα οποία μπορούν ακόμα να αναπαραχθούν αλλά έχει προέλθει... Δηλαδή από μια τέτοια κατάσταση απορρέει με μείωση. Και θα είχαμε για να χρησιμοποιήσω κοινή ορολογία κρίση. Περιβαλλοντική κρίση, λέει ο Και σε αυτά που λέγατε για τα συστημικά στοιχεία, θα είχαμε μειούμενο απόθεμα για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν θα είχε μόνο να κάνουν με την υπεραλίευση αλλά με την μόλυνση, με την κλιματική αλλαγή. Ε, προσπαθούμε λοιπόν υπό τις πολύ δύσκολες συνθήκες αυτές να εξασφαλίσουμε ότι το απόθεμα θα έχει την καλύτερη δυνατότητα αναπαραγωγής και ανανέωσης χωρίς να πάει σε καταστροφικές ε, μειωτικές τάσεις που θα οδηγούσαν στην ολική απαγόρευση. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ειδικά σε σχέση με αυτό, γιατί μιλάτε για εξαίρεση για ένα-δυο μήνες για τον γάδο, το οποίο μάλλον δεν ανταποκρίνεται στο πόσο καταστροφική η κατάσταση αυτή είναι, αλλά τι θα γίνει μετά. Όλα αυτά που αναφέρατε, τα περιβαλλοντικά, τη ρήπανση, όλα αυτά δεν θα εξαφανιστούν. Επομένως, θα κάνετε μετά, μετά την αναστολή για να βελτιωθεί συνολικά η κατάσταση για το γάδο. Okay. I mean, this goes slightly... Κοιτάξτε, αυτό ξεπερνάει λίγο τη μισθολογική μου κλίμακα που λέμε στα αμερικανικά. Αλλά κλιματική αλλαγή. Πρέπει κανείς να προσαρμοστεί σε αυτό και μάλιστα γρήγορα. Η IPCC θα δημοσιεύσει έκθεση για τις ε, παγωμένες ζώνες του πλανήτη το Σεπτέμβριο και γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζουμε από το σχέδιο, από το προσχέδιο, είναι ότι τα νέα δεν θα είναι καθόλου καλά. Η μείωση των, αποθέμα, των επαθεμάτων που μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα στη Βαλτική που είναι κλειστή θάλασσα. Είναι κάτι στο, προς το οποίο πρέπει να συνηθίσουμε. Είμαστε στο μέσον των αλλαγών αυτών των κλιματικών. Αν δείτε το προσχέδιο, θα δημοσιευθεί ξαναλέω το Σεπτέμβριο. Αλλά με ρωτάτε τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ σας λέω προσωπικά ότι πρέπει να επιγόντως, κατεπιγόντως να αναλάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα. το, τι, το πώς μπορούμε καλύτερα να διαχειριστούμε συνολικά τη Βαλτική θάλασσα με ξεπερνάει και πάλι την ειδικότητά μου και ίσως ξεπερνάει και την εντολή της Επιτροπής αυτής. Θα έπρεπε ίσως να συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Γεωργίας. Αλλά το φαινόμενο απαιτεί μια συστημική προσέγγιση. Εμείς με τα ε- έκτακτα αυτά μέτρα απλώς προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την πτυχή που αφορά τον αλλιευτικό πόρο. Αλλά σας ξαναλέω ότι η δραστηριότητα η αλλιευτική δεν είναι καν από μόνη της υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή. Υπάρχουν πολλά άλλα που θα έπρεπε να γίνουν για να αποτραπούν, αποτραπούν τέτοιες καταστροφές και τέτοια τραγωδία. Ε, ο πρόεδρος λέει αναφέρεται τόσο έτσι δραματικούς όρους και αναφέρεστε και στο απόθεμα του γάδου, εγώ δεν είμαι ειδικό, αλλά ξέρω ότι μέχρι να γίνει 7 ετών ηλικία ε, δεν έχει φτάσει σε, όριμο, σε όριμη ηλικία. Εάν εμείς όμως ε, ε, αλλιεύουμε γάδο πρωτού φτάσει σε αυτή την ηλικία, τότε γιατί δεν έχουμε αναλάβει μέτρα ήδη νωρίτερα. Ναι, έχετε δίκιο πρόεδρε. Ε, φτάνει σε ηλικία ορίμανσης αργά ο γάδος χρειάζεται να είναι σε μια αλφα ηλικία για να είναι πλήρω αναπαραγωγικό. Δεν αποκλείεται ότι μπορεί να αναπαραχθεί και νεαρότερο, αλλά όχι εξίσου συστηματικά, όχι εξίσου ομοιόμορφα ή αξιόπιστα. Στο παρελθόν έχουμε σε διάφορες περιπτώσεις μειώσει την ε, αλληλευτική ένταση και στην Ανατολική και στη Δυτική Βαλτική Ίσως να θυμάστε πριν από τρία χρόνια είχαμε μειώσει την ποσόστοση για το υπόλοιπο του βαλτικού γάδου 60% για να ευθυγραμμιστούμε σε μια έντονη πίεση συνολική. Και πέρυσι στο Συμβούλιο είχε γίνει αυτό. Θα γνωρίζετε ότι οι τελικές αποφάσεις για τα τάκ και τις για τις συνολικές δηλαδή επιτρεπτές ποσοστώσεις λαμβάνονται από το Συμβούλιο και όχι από την Κομισιόν, η Κομισιόν κάθε χρόνο υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με τι επιστημονικέ συμβουλέ. Και μερικέ φορέ το Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσει που αποκλίνουν για λόγους τους οποίους εγώ εδώ δεν πρόκειται να σχολιάσω. Αλλά από τις συμβουλές της ISIS αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η κυριότερη αιτία της μείωσης του αποθέματος δεν βρίσκεται στην, στο πεδίο της αλίας, αλλά σε άλλους παράγοντες, σε άλλες αιτίε που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό ευρύτερο τρόπο και με πολύ δύσκολο τρόπο. Η αλία είναι ένα μέσο διαχείριση που έχουμε, αλλά σίγουρα όχι το μόνο. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, σε ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος να παρατηρήσει κάτι, νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα αυτό και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν. Όταν μιλάτε για καταστροφή, τραγωδία, ε, ε, δεν θέλουμε να ξανααντιμετωπίσουμε τέτοια κατάσταση. Η Κομισιόν πρέπει εγκαίρως να κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και αν στο Συμβούλιο δεν λαμβάνονται οι απαραίτητε αποφάσεις εγκαίρως, εσείς πρέπει να μιλάτε ε, υψηλόφωνα, να ακούγεται η φωνή σα για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, και λέγοντας αυτά, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσία σας και την παρουσίασή σας. Yes, indeed. Um, right, um, uh, the next... Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την παράνομη λαθρεία και αναρχιαλία, την IUU, και επειδή δεν θέλουμε να μοιραστούμε με ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρουν ε, κάποια από τα μυστικά που θα συζητήσουν, θα ήθελα να ε, ζητήσω να αποχωρήσουν όλοι όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν, γιατί θα είναι και κλεισμένο των θυρών η συζήτηση, οπότε διακόπτουμε προσωρινά για 3-4 λεπτά.